Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε την συνεδρίασή μας. Εχθέ κάναμε τον πρώτο τριμερή διάλογο για το Erasmus for All και πριν έρθει ο κύριο Μαρτίνες θα ήθελα να σας ενημερώσω. Αν συμφωνείτε να κάνουμε αυτή την αλλαγή στην τριμερή διάταξη, εντάξει δεν υπάρχει αντίρρηση, ωραία. Σημείο 2 τη ημερήσιας διάταξη έγκριση των πρακτικών τη συνεδρίασης στις 18 Δεκεμβρίου. Αν υπάρχουν, ερωτι... αν υπάρχουν μέχρι το τέλος της ε, συνεδρίασης να τι πείτε για να τι συμπεριλάβουμε. Πάμε στο σημείο 3. Έχουμε ε, ε, διερμηνία σε όλες τις γλώσσες, εκτός από εστονικά, λιτονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα. Πρέπει επίσης να σας πω ότι 1η Μαρτίου ε, θα μας αφήσουν δύο συνεργάτες από τη γραμματεία. Η μία δεν θα πάει πολύ μακριά. Θα πάει στην Επιτροπή Τραν, η κυρία Κρισκάνε. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δουλειά που έκανε μέχρι τώρα. Όλοι όσοι έχετε δουλέψει μαζί της ξέρετε ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Την ευχαριστούμε λοιπόν και καλή επιτυχία στην Τραν. Θα είναι πολύ τυχερή που θα σας έχουν στη γραμματεία τους. Και μετά. Μετά από έξι χρόνια, δυστυχώς, πρέπει να σας ανακοινώσω. Όχι, δεν πεθαίνει. Η Ρίτα Σουάρες απλώς μας αφήνει και πάει στην Επιτροπή των Περιφερειών. Είναι... Θα είναι πια... Ήταν μάλλον το, το δώρο της Πρωτογαλίας σε εμάς και τώρα θα πάει στην Επιτροπή των Περιφερειών. Ε, δεν με ακούτε. Δεν με ακούτε καθόλου. Με θορύβους. Λοιπόν, για τον τρίλογο, στο το χθεσινό, ε, ήμουν εγώ, ήταν ο εισηγητής, ο σκιώδης εισηγητής, ε, ο κύριο Λόκεγκαρντ, η κυρία Μπατού, η κυρία Περζιάν δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι μαζί μας. Στην αρχή η πρόεδρος ε, η κυρία Άντερσεν είναι η πρόεδρος της ομάδας του Συμβουλίου, μας παρουσίασε την εντολή του Συμβουλίου και μας τόνισε ότι για την ίδια είναι πολύ σημαντικό και μας το έλεγε συνέχεια ξανά και ξανά να πλουστεύσουμε το κείμενο, να γίνει λίγο πιο συγκεκριμένο, αλλά το Συμβούλιο 1 τρίτο από τις ε, τροπολογίες μας ε, τις ε, δέχτηκε, που σημαίνει ότι υπάρχουν πολλά κοινά σημεία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Βεβαίω ε, είπαμε ότι υπάρχουν ε, ε, δυνατότητε να συζητήσουμε για το πού ακριβώς θα γίνει πιο συγκεκριμένο το κείμενο. Επίσης υπήρξε ένας κατάλογος τεχνικών αλλαγών που είχαμε συζητήσει και στην Επιτροπή μας, Τι είχαμε εγκρίνει ε, ήταν κυρίω λεκτικέ αλλαγέ, αν θα βάλουμε είτε, αν θα βάλουμε και, αν θα βάλουμε κάπου μια τελεία ή ένα κόμμα για να είναι πιο εύληπτο το κείμενο. Μετά, είχαμε δει αρκετά άρθρα για, όπου υπάρχουν διαφορέ μεταξύ του, των δύο θεσμικών οργάνων. Παρ' όλα αυτά οι διαφορέ μα ήταν μικρέ και έτσι προχωρήσαμε αρκετά. Τα σημεία τώρα στα οποία συμφωνήσαμε θα πρέπει το Συμβούλιο να τα συζητήσει στην ε, ομάδα εργασίας του και επειδή ακριβώς ε, ε, ήταν και οι σκιώδεις μαζί μας, ε, μπορέσαμε και εμείς να δώσουμε την απόψή μα. Τώρα, για την εποπτεία των αποτελεσμάτων και τη επίδοση. Άρθρο 17, πρόσβαση στα προγράμματα. Άρθρο 18, για τις χώρες μαζί με το εκτιμώντας 29α. Άρθρο 19, συμπληρωματικότητα μαζί με το εκτιμώντας 24. Ε, θέμα επίσης εθνικές αρχές, 22 εθνικοί οργανισμοί, εθνικές υπηρεσίες, 23 καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άρθρο 30 ε, επιτροπολογία και άρθρο 1 εύρος του προγράμματος και άρθρο 3 ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Υπάρχουν τρία σημεία τα οποία τα είπαμε ξεκάθαρα χτε, γιατί για μας είναι πολύ σημαντικά και ζητήσαμε από την Κομισιόν και το Συμβούλιο να τα σκεφτεί. Ένα θα σας αναφέρω γιατί υποθέτω ότι θα σας ενδιαφέρει η Επιτροπή Προγράμματος που είπαμε ότι ε, μια που είναι υπεύθυνη για όλα ουσιαστικά θα πρέπει να ε, έχει μια σύνθεση συγκεκριμένη όταν θα συνεδριάζει. Όταν μιλούμε για νεολαία θα πρέπει να, έχουν άνθρωποι, να είναι άνθρωποι εκεί που εκπροσωπούν τους νέους. Όταν μιλούμε για προγράμματα, για το κομμένιο Η κοινωνική σχετικοι επιρογνωμονες σε αυτη την επιτροπη η κοινωνικη μετερη τωρα θα προσκαλούνται ως ε, παρατηρητές. Αυτό ήταν μία από τις επιθυμίες μας και ήταν και η επιθυμία των πελατών μας ας πούμε. Το αναφέραμε στο Συμβούλιο, η Κομισιόν το κατάλαβε, το Συμβούλιο το κατάλαβε. Απλώς είπαν ότι αυτό είναι θέμα ιστορικού κανονισμού της Επιτροπής Προγραμματισμού. Και όταν, και όταν είπαμε ναι, αλλά αν δεν, ε, την, ε, αν δεν υπάρχει αυτό στον ιστορικό κανονισμό της Επιτροπής, πώς θα το διευθετήσει η Επιτροπή. Μας είπαν «Ε, εντάξει θα το σκεφτούμε, πώς μπορούμε με νομικό τρόπο να το προσθέσουμε στον ιστορικό κανονισμό. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο εμείς θεώρησαμε πολύ σημαντικό και που θα το ξανασυζητήσουμε. Κατά τα λοιπά, το κλίμα ήταν ιδιαίτερα θετικό. ήμασταν όλοι πολύ ευγενείς μεταξύ μα και υποθέτω ότι ε, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις. Η επόμενη ε, η επόμενη φορά που θα συναντηθούμε είναι 19 Μαρτίου. Νομίζω ότι αυτό πάει πολύ μακριά. Το Συμβούλιο σήμερα μας ρώτησε μήπως μπορούμε να κάνουμε ένα τριμερή διάλογο πιο νωρίς από τις 19 Μαρτίου. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε να το δρομολογήσουμε. Η Γραμματεία θα έρθει σε επαφή με την Γραμματεία του Συμβουλίου και θα παρακαλέσω και τους κοιόδης συγητές να συμβάλλουν. Ίσως θα μπορούσαμε να το δούμε στην επόμενη, ε, επόμενη εβδομάδα του Στρασβούργου. Ε, Ούτε ή άλλως όλοι εκεί θα είμαστε. Μπορούμε να κάτσουμε για μια μισή ώρα, δύο ώρες να, να το συζητήσουμε. Βέβαια, οι δύο ώρες δεν είναι και πολύ. Λοιπόν, αυτά από μένα. Πάμε στον, ε, στο σημείο 4. Να καλωσορίσω τον Μικελάνχελ Μαρτίνες Μαρτίνες. Είναι ο πρόεδρος της ομάδας επαφής του Προεδρείου για το σχέδιο για το σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Δεν θέλω να προσθέσω τίποτα, τον έχουμε ήδη δύο φορές προσκαλέσει εδώ και θέλω να, μας, να του δώσουμε τον, τον λόγο για να μας μιλήσει. Η κυρία Παλιαδέλη είναι μέλος επίσης αυτής της ομάδας, έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να εκπροσωπείται πάντα. Και υπάρχουν και δύο παλιοί συνάδελφοι εδώ, ο κύριος Ωνεστά και ο κύριος Βίρτς, οι οποίοι επίσης ενδιαφέρονται για το θέμα. Είναι, είμαστε καλή ομάδα λοιπόν και έχουμε προχωρήσει αρκετά. Τώρα πόσο έχουμε προχωρήσει συγκεκριμένα θα μας πει ο καλός μας φίλος Μικελ Άγχελ. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητή Ντόρις. Πράγματι, αποτελεί μεγάλη ικανοποίηση το γεγονός ότι είμαι εδώ ενώπιον της Επιτροπής σας να μιλήσω για το σχέδιο αυτό και πρόκειται για κάτι το οποίο γνωρίζουν πολλοί από εσά. Εδώ δίπλα μου είναι η κυρία Ρέα Βαγκάλη, η οποία είναι η διευθύντρια της ομάδος που προχωρά τις εργασίες ε, του σχεδίου αυτού. Όπως ε, έλεγε και η πρόεδρος, έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές. Είναι η έκτη φορά που ερχόμαστε εδώ ενώπιον της Επιτροπής, την τέταρτη φορά ε, σε αυτή τη θητεία και θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι από το Δεκέμβριο το Δεκέμβριο του 2008 η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας ενέκρινε ήδη ε, ένα βασικό κείμενο το οποίο είχε εκπονήσει μια ομάδα ε, εγνωσμένου κύρους εμπειρογνωμόνων σε θέματα ιστορίας και μουσιολογίας. Και θα ήθελα εδώ να σταθώ σε κάτι το οποίο είπε η Ντόρις το γεγονός ότι τόσο η πρόεδρος της Επιτροπής όσο και η κυρία Παλιαδέλη εργάστηκαν με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο και με ενθουσιασμό για το σχέδιο αυτό και θα πρέπει να τις ευχαριστήσουμε ε, βάθους καρδίας ε, για το γεγονός ότι ενδιαφέρθηκαν τόσο πολύ για το θέμα αλλά και για την ε, ε, διάθεσή τους να εργαστούν διότι πρόκειται για ένα ζωντανό πρόγραμμα το οποίο προχωρά και διαμορφώνεται όσο προχωράει και το να έχουμε στην ομάδα μας δύο συναδέλφους που βοηθούν τόσο πολύ το πρόγραμμα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δράτομαι δε και της ευκαιρίας ε, για να σας εξηγήσω τι ακριβώς έχει γίνει, πώς έχουν προχωρήσει τα πράγματα σε ένα χρόνο, δεδομένου ότι την τελευταία φορά που ήμουν εδώ ήταν 29 Φεβρουαρίου. 29 Φεβρουαρίου πέφτει σε δίσεκτο έτους, μια φορά κάθε τέσσερα χρόνια. Επομένως, ε, τότε ε, συναντηθήκαμε τελευταία φορά για να δούμε λίγο πώς προχωράει το όλο πρόγραμμα. Θα σας πω λοιπόν τι πρόοδος έχει επιτευχθεί, ε, τι γίνεται στο κτίριο και τι γίνεται όσον αφορά το περιεχόμενο του προγράμματος, ε, τις έρευνες που έχουν γίνει για τις ε, δυνατότητες επισκέψεων, την, ε, τον προγραμματισμό και ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει ε, εμένα και θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας αφορά την διάσκεψη που προβλέπετε λόγω του προγράμματος και επίσης και κάποια σχόλια για τον προϋπολογισμό. Να δούμε λοιπόν και τι γίνεται με αυτή τη διάσταση, η οποία λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες ήταν ένα από τα πιο ε, ταραγμένα, αν θέλετε, ζητήματα. Όσον αφορά το περιεχόμενο, θα πρέπει να πούμε ότι ο χώρος για τη μόνιμη έκθεση του ε, κτηρίου Eastman, το οποίο γνωρίζετε νομίζω όλοι που βρίσκεται, είναι εδώ πίσω στο πάρκο Λεοπόλντ, ε, λίγα μέτρα από το κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η μόνιμη έκθεση λοιπόν, ε, η οποία θα βρίσκεται, θα στεγάζεται στο κτίριο Eastman, βρίσκεται στους πέντε ε, ανώτερους ορόφους, ενώ στους δύο πρώτους ορόφους ε, έχουμε διατηρήσει το χώρο για προσωρινές εκθέσεις η ομάδα από τότε που ξεκίνησε να εργάζεται στις αρχές του 2011 και το καλοκαίρι ε, το περασμένο κατάφερε να καθορίσει ποιο θα είναι το πνεύμα της μόνιμης έκθεσης. Ε, αυτό το οποίο ετοιμάζουν οι φίλοι μας ε, υπό την διεύθυνση της Τάγια είναι ακριβώς το τι ακριβώς θα περιλαμβάνει αυτή η μόνιμη έκθεση. Ε, να δούμε ποια περίοδο θα καλύπτει η μόνιμη έκθεση και τι θεματικές ενότητες θα έχουμε στην έκθεση. Βασιζόμαστε φυσικά στο βασικό έγγραφο το νεολογικό που ετοιμάσαμε το 2008 και το οποίο εξελίχθηκε με τη βοήθεια ε, του σχεδιαστή. Έχουμε κάποιες εικόνες που έχουμε στην συνεδρίαση. Ε, αυτές είναι από τον αρχιτέκτονα και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι από τότε που έγινε η πρόσκληση ε, προτάσεων για τον διαγωνισμό και τη διαδικασία επιλογής της επιχείρησης που θα κάνει τον τελικό σχεδιασμό για την τελική έκθεση έχουμε προχωρήσει. Ε, στο Προεδρείο του Κοινοβουλίου υποβλήθηκε ε, ένα σχέδιο και εγκρίθηκε την 1η Οκτωβρίου του 2012 και ε, έχει ως εξής. Έχουμε την ευρωπαϊκή ιστορία του 20ου αιώνα που θα είναι ο βασικός πυρήνας της μόνιμης έκθεσης και λίγο πολύ θα είναι το 75% της διαθέσιμης επιφάνειας της έκθεσης και θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ε, όπως έχει ξεκινήσει μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου ε, Αιώνα, λαμβάνοντας υπόψη και το τι συνέβη στο Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο. Ε, το δεύτερο τμήμα της μόνιμης έκθεσης, το οποίο θα είναι μικρότερης έκτασης ε, και θα είναι και ένα τμήμα του δεύτερου ορόφου της ε, μόνιμης έκθεσης, θα έχουμε ε, τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σε προηγούμενους αιώνες ε, και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε για να κατανοήσουμε τι συνέβη στον 20ο αιώνα. Είναι δηλαδή γεγονότα τα οποία είχαν μεγάλη σημασία και πάντα οι ιστορικοί που ασχολούνται με το θέμα έλεγαν ότι δεν θα πρέπει να τα παραγνωρίσουμε και εγώ νομίζω ότι ενώ θα έπρεπε να επικεντρωθούμε κυρίως στο τι συμβαίνει στον 20ο και στον 21ο αιώνα, αλλά οι ιστορικοί που συνεργάζονται μαζί μας επιμένουν ότι υπάρχουν κάποια γεγονότα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για να κατανοήσουμε τι συνέβη στον 20ο αιώνα. Ιδίω το δεύτερο μισό του 20 ο αιώνα θα πρέπει λοιπόν να είναι σαφή κάποια σημεία αναφοράς τα οποία ε, έχουν γίνει πολύ πιο πριν. Το δεύτερο τμήμα στο δεύτερο όροφο της έκθεσης θα είναι αφιερωμένη κυρίως στους δύο παγκοσμίους πολέμους, τον πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και από τον τρίτο όροφο και πέρα έχουμε την η πολιτική ιστορία της Ευρώπης που θα συμπληρωθεί με οικονομικές, κοινωνικές, ε, πολιτισμικές και προσωπικές πτυχές. Στον ε, τέταρτο και πέμπτο, τρίτο και τέταρτο όροφο θα πάμε από το 1945 μέχρι τις μέρες μας και θα δούμε τι γίνεται και με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της ευρύτερης ευρωπαϊκής ιστορίας, δηλαδή και κάποιες αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει σε περιοχές της Ευρώπης που δεν ήταν ή που δεν ε, είναι τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον πέμπτο όροφο θα έχουμε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο, θα είναι πιο διαδραστική η επικοινωνία και θα υπάρχει μια συζήτηση για τις ε, ε, παρούσες προκλήσεις και τις μελλοντικές προκλήσεις. Ε, η έγκριση του Προεδρείου δόθηκε και από εκεί και πέρα η ακαδημαϊκή ομάδα ετοιμάζει διάφορα στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν να αφηγηθούμε την ιστορία την οποία θα περιγράφουμε στη μόνιμη έκθεση. Ε, είναι και η επιχείρηση που ασχολείται με το σχεδιασμό ε, αυτή η οποία θα μας βοηθήσει και ελπίζω να καταλήξουμε σε μία έκθεση η οποία κατά την άποψή μου θα υποδηλώνει πολλά και ε, η ομάδα που εργάζεται υπό τη διεύθυνση της ΤΑΙΕ η οποία μας έχει δώσει αρκετές αποδείξεις ότι έχει εξαιρετικέ δυνατότητες, ε, θα μας δώσει το τελικό αποτέλεσμα. Δεν θα σας ε, κρύψω βέβαια ότι από τη δική μας την πολιτική εμπειρία το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο, έχει πάρα πολλέ δυσκολίες όσοι είχαμε την τύχη να γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πώς έχει προχωρήσει όλη η διαδικασία της ιστορίας του οίκου, της γερμανικής ιστορίας και των ε, ε μουσείων της Βόνης και του Μουσείου του, της Λιψίας, εδώ έχουμε την ίδια διαδικασία, πολλαπλασιασμένη επί 27, διότι τόσα είναι τα κράτη-μέλη που επηρεάζουν το συγκεκριμένο μουσείο και φυσικά ε, το ενδιαφέρον που δείχνουν διάφοροι για το θέμα. Ε, πρέπει να σας πω ότι εγώ συναντήθηκα πολύ περισσότερες φορές με τον πρέσβη της Ρωσίας και τον πρέσβη της Τουρκίας από ότι με τους πρέσβεις των χωρών μελών της Ένωσης, διότι φυσικά και η ΜΕΝ και η ΔΕ ανησυχούν για το όρομα το οποίο θα παρουσιάσουμε για την Ευρώπη, πώς θα την παρουσιάσουμε την Ευρώπη και πώς θα παρουσιάσουμε το ρόλο που διαδραμάτισε η Ρωσία, η Σοβιετική Ένωση, η Τουρκία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η πιο σύγχρονη Τουρκία στο, είναι όλη αυτή διαδικασία και εμείς θέλουμε φυσικά να την περιγράψουμε και φυσικά δεν μπορούμε να την ε, αντιληφθούμε εντός ε, στενών πλαισίων, στενών ορίων, λησμονώντας ε, σημαντικούς καθοριστικούς παράγοντες για κάποια γεγονότα της ιστορίας των χωρών μας και συμπεριλαμβάνει και της ιστορίας της διαδικασίας που μας έχει οδηγήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. τώρα, για να περάσουμε τώρα στη συλλογή. Η συλλογή που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε έχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια σημαντική συλλογή μουσείου ξεκινώντας από το μηδέν. Και με αυτή την προοπτική, με αυτό το πρίσμα, η Ακαδημιακή Ομάδα του Προγράμματος καθόρισε μια πολιτική για το τι θα γίνεται με τις συλλογές και καθόρισε τα βασικά κριτήρια επί των οποίων θα ε, αποκτήσουμε ή θα ζητήσουμε ε, για δανεισμό και θα μας δοθούν συγκεκριμένα αντικείμενα για τη συλλογή. Ε, έτσι γίνεται συνήθως για να έχουμε μία συλλογή. Θα πρέπει να υπάρχει και ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης της συλλογής από εκεί και πέρα και ε, ένα πλαίσιο βάσει των οποίων θα μπορούμε να δούμε τι γίνεται με τη συντήρηση ε, των ε, αντικειμένων και θα πρέπει να γίνεται με σύγχρονο και επαγγελματικό τρόπο. Ε, πρόσφατα είχαμε ένα πολύ σημαντικό βήμα, διότι ξεκινήσαμε με κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. ουσιαστικά την ταυτότητα της, του προγράμματός μας. το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησαν το μετάλλιο και το πιστοποιητικό του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης ε, να ε, βρίσκονται στο ε, νίκο της ευρωπαϊκής ιστορίας. Αυτή η είδηση είχε μεγάλη σημασία σε όλες τις χώρες μας και πρέπει να σας πω ότι ευτυχώς λόγω της ε, ανακοίνωσης ότι το μετάλλιο και το βραβείο Νόμπελ θα βρίσκονται στον οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, υπήρξαν πάρα πολλές διαβουλεύσεις, ε, μας ρώτησαν πάρα πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης για το πρόγραμμα που μέχρι τώρα δεν ήξεραν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο στα σκαριά και δώσαμε, έτσι, μας δόθηκε η δυνατότητα να τους εξηγήσουμε λίγα πράγματα. Πέραν αυτών των αντικειμένων έχουμε ήδη και πάνω από 70 αντικείμενα από τις διάφορες τελετές ε, που έγιναν στη Όσλο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τεκμηριώσουμε όλες αυτές τις τελετές για το Νόμπελ Ειρήνης, όχι μόνο το δικό μας το Νόμπελ που δόθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ε, άλλα Νόμπελ τα οποία θα μπορούσαν ίσως να έχουν σχέση με την πρόσφατη ιστορία της Επίρου μας. Αυτό ήταν το πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο κατέδειξε πόσο σημαντικό είναι να ε, έχουμε ένα θεσμό ο οποίο προσπαθεί να διατηρήσει ε, αντικείμενα που καταδεικνύουν πώ ε, διαμορφώθηκε η ιστορία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ειπα επιση επίσης ότι υπήρχαν ένα-δυο πράγματα τα οποία θα έπρεπε να σχολιάσουμε. Ε, καταρχάς, οι σφιγμομετρήσεις. Η ακαδημιακή ομάδα στη διάρκεια του προηγουμένου έτους έκανε μια πρώτη σειρά από σφιγμομετρήσει για πιθανού επισκέπτε να δούμε κατά πόσο πόσον γνωρίζουν και κατά πόσον έχει ενδιαφέρον το κοινό ε, να έρθει να δει την έκθεση στο μέλλον και για να προσαρμόσουμε και την έκθεση ε, ανάλογα με διάφορα στοιχεία τα οποία θα ανακύψουν από τις ε, έρευνες αυτές. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ιδίω για όσου επισκεπτόμαστε πάρα πολλά μουσεία για να δούμε πώ λειτουργούν τα πράγματα, ότι το μουσείο μα θα έχει ένα προνόμιο σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα μουσεία που έχουμε επισκεφθεί οποιοδήποτε άλλο μουσείο ανοίγει, η πρώτη ανησυχία του ομάδα που το διευθύνει είναι πώ θα προσελκύσει το ευρύ κοινό. Εμεί έχουμε το προνόμιο να ανοίγουμε ένα μουσείο με ένα εκατομμύριο επισκέπτε που θα περιμένουν στην ουρά. Ε, ή με ένα εκατομμύριο δυνητικού επισκέπτε που θα περιμένουν στην ουρά, διότι όλε οι ομάδε που μα επισκέπτονται, όλοι όσοι πλησιάζουν εδώ στην περιοχή, σίγουρα στο πρόγραμμά του θα περιλαμβάνεται και η επίσκεψη στον οίκο τη Ευρωπαϊκή Ιστορία. Και κάτι το οποίο προέκυψε και είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχει και μια ομάδα επικοινωνίας και στην ε, διοικητική πρωτοβουλία της, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, συμπεριλήφθηκε και στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ε, το θέμα και νομίζω ότι αυτό μας βοηθάει ιδιαίτερα. Θα ολοκληρώσω με ένα λεπτό ζήτημα το οποίο θα ήθελα να σας παρουσιάσω με πάσα προσοχή, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Στις 9 Μαΐου φέτος, στο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατόπιν παρακίνηση του Προέδρου μας, Ο πρόεδρος είπε ότι ίσως θα έπρεπε να γίνει μια μεγάλη διάσκεψη με προσωπικότητες από τον χώρο των μουσείων της ιστορίας, ε, θεούς και ανθρώπους, ώστε κατά κάποιο τρόπο να ανακηρύξουμε, να, να, να δηλώσουμε στον κόσμο το πρόγραμμα αυτό και πώς προχωράει. Ε, προχωρούμε αυτή την ιδέα και η αλήθεια είναι ότι διάφοροι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, η Επιστημινική Επιτροπή και κάποιοι άλλοι, διαπιστώσαμε ότι αυτή η μεγάλη διάσκεψη θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμη, αλλά θα μπορούσε ίσως να δημιουργήσει και αρκετά προβλήματα, ιδίω εάν δεν οργανωθεί από την ίδια ομάδα που ε, προχωρά το πρόγραμμα. Δεν σας κρύβω ότι στο χώρο των μουσείων και της ιστορίας ε, ερίζουν οι απόψεις και υπάρχει και μεγάλος φθόνος, ε, αρκετές επικρίσεις και αυτό το οποίο ελοχεύει ως κινδύνος είναι αυτή η μεγάλη ε, διάσκεψη που θα είναι τα εγγένεια ουσιαστικά στην πραγματικότητα θα μπορούσε να δυναμητήσει το πρόγραμμα ή να δημιουργηθεί σωρία επικρίσεων από διάφορες πλευρές και να γίνει ουσιαστικά είναι από ο τάφος μας αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων θα μπορούσε να καταλήξει πάρα πολύ άσχημα. Δεν θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να πυρπολίσουμε μια τόσο ε, ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία και να θεωρήσουν ότι είναι σκάνδαλο, διότι ξέρετε ότι υπάρχουν μέσα μαζική ενημέρωση που είναι κατά του προγράμματο και άνθρωποι που είναι κατά του προγράμματο, κάποιοι γιατί είναι κατά τη Ευρώπη και είναι αντίθετοι σε κάτι τέτοιο και κάποιοι άλλοι γιατί θεωρούν ότι δεν θα έπρεπε να έχει αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευτυχώ έχουμε ήδη πείσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και θα συμμετέχει στην ε, συντήρηση ε, του μουσείου όταν θα ξεκινήσει η λειτουργία του. Ε, θα πρέπει παρόλα αυτά να πούμε ότι η ημερομηνία για αυτή την διάσκεψη ε, ακόμα δεν έχει ε, καθοριστεί. Όλοι θεωρούμε ότι θα πρέπει να καθυστερήσει όσο το δυνατόν περισσότερο για να γίνει όταν θα έχουν πλέον εδρεωθεί τα πάντα. Κάτι τελευταίο το οποίο θα ήθελα να σας πω είναι ότι ο προϋπολογισμός προχωρά λογικά. Το Προεδρείο το Σεπτέμβριο του 2011 ενέκρινε ένα προϋπολογισμό 6,4 εκατομμυρίων ευρώ και αυτό το οποίο αποφάσισε το Προεδρείο με την Επιτροπή Προϋπολογισμών που ξέρετε ότι σε αυτή την περίπτωση διατάζει ότι αντί να το εγγενιάσουμε το 2014 όπως είχε προβλεφθεί, θα το εγγενιάσουμε το 2015 ή το 2016, ώστε τα τελικά ποσά τα οποία έχουν διατεθεί για το πρόγραμμα να μπορέσουν να, να επεκταθούν και έτσι να κατανεμηθούν σε διάφορα έτη προπολογισμού. Αυτά είχα να σας πω. Ε, σας ευχαριστώ όπως πάντα για την προσοχή σας και να επαναλάβω ε, για άλλη μια φορά ότι όπως πάντα είμαι στη διάθεσή σας για το επόμενο τέταρτο περίπου ώστε να ακούσω τις απόψεις σας και να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση ή οποιοδήποτε σχόλιο θέλετε να κάνετε. Ευχαριστώ Ντόρι. Ε, Εγώ ευχαριστώ Μιγέλ. Δύο έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Καβαντά πρώτα. Je vous remercie. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Μιγγέλ για την αυτή ενημέρωση. Θα ήθελα να διευκρινίσουμε δύο-τρία πράγματα επί τη ευκαιρία αυτής της παρουσίασης. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ξεκάθαρα ότι η Ευρώπη αξίζει τη μνήμη και μάλιστα αποτελεί αυτό υψηλή αναγκαιότητα. Δεν μιλώ για εθνικέ μνήμε, μέσα δηλαδή στα κράτη-μέλη, αλλά μια κοινοτική μνήμη. Κάτι το οποίο ακόμη δεν υπάρχει με μια πρακτική υλική ε, μορφή με ένα τέτοιο κτίριο δηλαδή. Γι' αυτό και η ιδέα του μουσείου είναι πραγματικά ευπρόσδεκτη. Θα ήθελα επίσης να πω ότι δεν καταλαβαίνω ούτε και δέχομαι αυτή την αντιπαράθεση που λέει ότι ίσως το κοινοβούλιο δεν είναι το όργανο που και τα λοιπά. Όχι, ακριβώς το αντίθετο ισχύει. Αν υπάρχει ένα όργανο που θα έπρεπε να το κάνει είναι το όργανο που απαρτίζεται από τους αιρετούς εκπροσώπους ε, των λαών της Ευρώπης. Δεν μπορούμε να ε, περιοριστούμε και να ε, δείχνουμε ένα πρόσωπο της Ευρώπης που χαρακτηρίζεται από μια τεχνοκρατική αοριστία. Το κοινοβούλιο είναι αυτό το οποίο πρέπει να λάβει την αποστολή και ε, θα πρέπει να ε, έχουμε αυτό το μουσείο το οποίο θα είναι αφιερωμένο στην κοινοτική μνήμη και θα λάβω την ε, πρωτοβουλία, αν συνεχιστούν όλες αυτές οι διαμαρτυρίες, ε, να, συνεχί... να κάνουμε μία αναφορά στο διαδίκτυο για να συλλέξουμε υπογραφές, διότι δεν είναι δυνατό να υπάρχουν αυτές οι επιφυλάξεις που, εντάξει, για τις οικονομικές δυσκολίες το καταλαβαίνω και υπάρχουν. Ε, είναι λίγο λεπτό το θέμα και αυτό ισχύει παντού και για όλα τα δημιουργήματα που φυλάσσουν την ιστορική μνήμη και για πολλά ιστορικά κτίρια υπάρχουν ζητήματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να φοβόμαστε το αντίθετο. Πρέπει να, ε, πραγματικά να κάνουμε ακουστεί η φωνή μας για να στηρίξουμε αυτό το project. Αυτή είναι η πρώτη μου σκέψη. Θα ήθελα επίσης να πω ότι οι πρόεδροι των ομάδων που ουσιαστικά αποτελούν την κατευθυντήρια γραμμή, θα έλεγα, στο Κοινοβούλιο, τις μείζονες ομάδες αναφέρομαι, θα πρέπει να φροντίσουν ε, η κομματική πολιτική να υποκληθεί, θα έλεγα, μπροστά στο σεβασμό της ιστορικής μνήμης της Ευρώπης και των επιτυχιών της, αλλά και των αποτυχιών της. Είχαμε στιγμές μεγάλης ευημερία και είχαμε και πολλές τραγωδίες. Βιώσαμε τέτοιες και φέτος και πέρυσι. Αλλά πρέπει να διδαχθούμε από όλα αυτά. Και η οικοδόμηση, η ανέγερση αυτού του μνημείου σε καμία περίπτωση άλλωστε δεν είναι ε, φαραωνική, δεν ε, είναι μεγαλόσχημα αυτά τα οποία θέλουμε να πετύχουμε. Θα έλεγα μάλιστα ότι ο προεπολισμός είναι και μετριοπαθής. Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, αγαπητέ Μιγγέλ, είναι η στεναρή, η θαραλέα απάντηση ε, για όλους αυτούς τους πολέμους που θα παραμείνουν ε, ανεξίτηλα γραμμένοι στη μνήμη όχι μόνο των γενιών που έχουν προηγηθεί, των σημερινών, αλλά και των πολλών ακόμα μελλοντικών γενιών. Δεν θα πρέπει λοιπόν ε, να παραβλέπουμε. Σίγουρα υπάρχουν επιστήμονες πάρα πολύ φωτισμένοι. Από τη στιγμή που λένε λοιπόν ότι πρέπει να περιλαμβάνονται και κάποια άλλα γεγονότα, νομίζω ότι θα πρέπει να τα συμπεριλάβουμε γιατί αυτά μας ε, ε, καθορίζουν, καθορίζουν τον, το από πού προερχόμαστε και το τι είμαστε σήμερα. Επίσης, αρκεί να δει κανείς τι γίνεται σήμερα στις χώρες, ε, το ρεβισιονισμό που βλέπουμε να σημειώνει αύξηση, τις τεράστιες δυσκολίες γενικά που αντιμετωπίζουμε. Μία φράση του Λιβιζέλ ως ε, προειδοποίηση και για το μέλλον θέλω να σας υπενθυμίσω και που μας είχε πει Ευχαριστώ για τα 60 χρόνια, αλλά μην ε, ε, χαλαρώσετε τις πιέσεις. Αυτό ήταν στο βραβείο Νόμπελ και ο Ελί είχε πει ότι οι λαοί που δεν γνωρίζουν την ιστορία τους ε, είναι εκτεθειμένοι και θα χρειαστεί να την ξαναζήσουν την ιστορία τους. Και αυτό, αυτή τη ρίση του Ελί τη συμμερίζομαι 100%. Αυτός ο κίνδυνος υπάρχει και στην περίοδο της ειρήνης, πόσο μάλλον θα έλεγα. Και όλα αυτά τα θέματα βέβαια κάτι που δεν αναφέρθηκε, θέλω να προτείνω εδώ, μάλλον αναφέρω, είναι μια πρόταση. Όλα αυτά λοιπόν έχουν και μια πρόταση για βιογραφίες ε, ή για πορτρέτα κάποιων ανθρώπων που έδωσαν τη ζωή τους για δύο διαδοχικές ε, τυραννίες. Αγωνιζόμουν κατά δύο διαδοχικών τυραννιών. Την ναζιστική τυραννία βέβαια, αλλά και κάτι που ίσως είναι πιο δύσκολο, αλλά είναι κάτι πολύ σημαντικό και πρέπει να το πούμε, είναι η Σοβιετική τυραννία που εχμαλώτησε ε, χώρες, ε, λαούς που σήμερα είναι εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί μας. Δεν μιλάω με βάση την ιδεολογία μου, δεν κάνω ιδεολογική συζήτηση εδώ. Σας καλώ να εγκύψετε σε βιογραφίες κάποιες θα τις βρείτε στα γερμανικά, στα αγγλικά, ε, βιογραφίες ανθρώπων που δεν τους γνωρίζουμε, ιδίως εδώ στην ε, Δύση, κυρία Γκούζη Φλάσμαν για παράδειγμα στην Πρατισλάβα, ο κύριος Ζέλ Μπραντ στην ε, Βουδαπέστη, ο σύμβαλος Ραούλ, σύμβουλος Ραούλ Βάλεμπεργκ και πάρα πολλοί άλλοι. Αυτοί οι άντρες, αυτές οι γυναίκες που ανήκουν στην σύγχρονη μνήμη, στη μνήμη του 21ου αιώνα που μιλούν για αντίσταση, ε, που έχουν μεταλαμπαδεύσει το, το πνεύμα της αντίστασης. Νομίζω ότι αξίζουν αυτοί οι άνθρωποι όταν μπαίνει κανείς στο μουσείο ή οπουδήποτε αλλού κρίνεται στη μου, αξίζει να φαίνονται να είναι αυτό το μονοπάτι ε, της ειρήνης ε, μία, αν θέλετε, γαλαρία με τα προτρέτα τους. Πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους θυμόμαστε. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, κυρία Τρούπελ. Ευχαριστώ. Γενικώ ε, συμμερίζομαι με την άποψη που λέει ότι δεν έχουμε μόνο ανάγκη για αθνική μνήμη, αλλά και για μια κοινή ευρωπαϊκή ε, μνήμη που προκύπτει από την πολυσχηδή ιστορία της ε, Ευρώπης. Μιλούμε για πολύ πλούσια ιστορία, για πολύ διαφορετική. Και το σημαντικό είναι, και το έχω ξαναπεί όταν μιλούσαμε για, την, για τον οίκο αυτό της ευρωπαϊκής ιστορίας, ότι πρέπει να συνεργαστούμε και να συνδυάσουμε και τα υπάρχοντα μουσεία που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ας πούμε υπάρχει το Μουσείο Κατοχής στην Ρήγα και το Μουσείο που αφορά τους βασανισμούς στη Βουδαπέστη. Νομίζω ότι όλα αυτά τα μουσεία θα πρέπει να συνδυαστούν με κάποιο τρόπο, έτσι ώστε να ξέρουν ότι εδώ υπάρχει ένας οίκος για τους Ευρωπαίους πολίτες, έτσι ώστε να, να μπορούν να έρθουν και εδώ και βεβαίως να το γνωρίζουν. Και ένα τελευταίο για τον προπολογισμό. Έχουμε το αποτέλεσμα της έκτακτη ε, συνόδου κορυφής για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο με μείωση των διοικητικών δαπανών. Έχετε συζητήσει στο Προεδρείο του Κοινοβουλίου αν υπάρχει οποιαδήποτε συνέπεια ε, αυτή της τη απόφαση στο ε, προπολογισμό για το σπίτι τη Ευρωπαϊκή Ιστορία. Θα ήθελα να μου το πείτε, γιατί για μένα δεν είναι απόλυτα σαφέ αν, αν, υπάρχει αντίκτυπο ή όχι. Ο κύριο Ταβάρε.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 καθηγητές μου της ιστορίας έλεγε ότι όταν θυμόμαστε την ιστορία μας πρέπει να θυμόμαστε ότι οι άνθρωποι που έκαναν τα λάθη ή οδηγήθηκαν σε τραγωδίες δεν ήταν πιο ανόητοι από εμάς. Ας μην είμαστε λοιπόν κι εμείς πολύ περήφανοι και ας μην θεωρούμε ότι είμαστε πολύ πιο έξυπνοι από τους ε, παλαιότερους. Ας μην θεωρούμε ότι δεν μπορούν να ξανασυμβούν αυτά που έχουν συμβεί πριν από 100 ή πριν από 200 χρόνια ή άλλα πράγματα που έχουν ε, γίνει ε, ακόμα και πολύ πιο πρόσφατα, ακόμα και μετά τον ε, Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θεωρούμε ότι ήταν εξαιρετικοί διπλωμάτες, εξαιρετικοί πολιτικοί εκείνης της εποχής και εμεί ε, είμαστε, θεωρούμε ότι είμαστε ανώτεροι από αυτού, ότι είμαστε πιο έξυπνοι, πιο ικανοί. Όχι, θα πρέπει να είμαστε πιο συντηρητικοί, πιο ταπεινοί. Ούτε εμεί είμαστε τέλειοι, ποτέ δεν θα υπάρξει τέλεια ιστορία. Η ιστορία ποτέ δεν θα είναι 100% ουδέτερη. Θα είναι πάντα μια ιστορία την οποία θα πρέπει να δεχτούμε έτσι όπω είναι. Έχω να θέσω ένα ερώτημα. Το πρόβλημα αυτό με αυτή τη μεγάλη διάσκεψη, πώς θα το λύσουμε. και σε σχέση και με τις εκθέσεις που θέλουμε να περιλαμβάνονται στο μουσείο. Μιλούμε για διαχείριση του παρελθόντος και σίγουρα ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος ε, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ε, είναι ένας πόλεμος που δεν τον κατάλαβε ποτέ κανείς 100%. Αλλά ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος προκάλεσε το δεύτερο. Και νομίζω ότι όταν μιλούμε για το παρελθόν, όταν σκεφτόμαστε το παρελθόν, συνήθως σκεφτόμαστε περισσότερο τον πρώτο παρά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Γι' αυτό νομίζω ότι εφόσον θα ανοίξουμε αυτό το μουσείο, εφόσον θα έχουμε αυτό τον οίκο της ευρωπαϊκής ιστορίας, το 2014 θα πρέπει να κάνουμε ίσως ένα συμπόζιο ένα, μια μεγάλη διάσκεψη και να, την, να, το σκεφτούμε πάρα πολύ προσεκτικά. Επιμένω στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο γιατί ήταν πραγματικά ένα τεράστιο γεγονός και είχε και τραγικές, τραγικές συνέπειες για τον 20ο αιώνα. Αλλά δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο τις τραγωδίες και μόνο τις άσχημες στιγμές. Γι' αυτό θα ήταν καλό ίσως στο μέλλον να υπάρξει ίσως μια έκθεση που θα δείχνει το μέλλον του παρελθόντος, ας πούμε τον ε, ε, Βίκτορ Ουγκό, τον Σπινέλη ε, και ανθρώπους δηλαδή που σκέφτηκαν για το μέλλον της Ευρώπης και πώς αυτό θα δομηθεί και που προσπάθησαν να αποφύγουν διάφορες τραγωδίες ή να αποτρέψουν διάφορες τραγωδίες που τελικά συνέβησαν. Είναι λοιπόν ένα μουσείο του μέλλοντος του παρελθόντος. Μιλούμε για το τρέχον ε, παρελθόν πολλές φορές. Εγώ τώρα σας προτείνω να σκεφτούμε το μέλλον του παρελθόντος. Και επίσης για τα εθνικά μουσεία. Ε, είναι καλή ιδέα να τα συνδυάσουμε. Ε, το είπε η κυρία Τρούπελ, υπάρχουν πολλά μουσεία που μπορεί να θέλουν να οργανώσουν κάποιες εκθέσεις στον δικό μας οίκο ιστορίας. Ας πούμε το Μουσείο Μετανάστευσης. Και στη Βραζιλία υπάρχει και στη ΣΥΠΑ εκεί ε, η, η, μετανάστευση και όλα τα έργα που υπάρχουν εκεί ε, προέρχονται από Ευρωπαίους που μετανάστευσαν στους χώρες, στις χώρες αυτές. Οπότε ίσως να μας ενδιαφέρει και εμάς να δούμε πώς ε, κινήθηκε η τάση αυτή. Να συνδυαστούν λοιπόν τα εκθέματα από τα διάφορα εθνικά μουσεία και βεβαίως και τα δικά μας τα εκθέματα θα μπορούσαν ίσως να εκτεθούν σε άλλες εκθέσεις Όχι μόνο να προσκαλούμε μουσεία εδώ, αλλά να πηγαίνουμε και εμείς εκεί. Οπότε αυτά τα εκθέματα δεν χρειάζεται να παραμένουν μόνο στην, ε, στις Βρυξέλλες, θα μπορούσαν όντως να ταξιδεύουν ουσιαστικά από ε, πόλη σε πόλη. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ο Μιγγέλ σε πέντε λεπτά πρέπει να φύγει, οπότε θέλει να απαντήσει τώρα και μετά ούτως ή άλλως θα μας μιλήσει η υπεύθυνη των ε, εκθέσεων για τα υπόλοιπα ερωτήματα εφόσον υπάρξουν. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ όσους πήραν το λόγο. Ε, πέντε λεπτά έχεις, Μιγέλ, παρακαλώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Ντόρις. Πράγματι, δυστυχώ πρέπει να φύγω γιατί έχω μια πτήση να προλάβω. Αλλά η Διευθύντρια σίγουρα θα απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα. Θα ήθελα να απαντήσω σε δύο σχόλια βέβαια, σε όσα είπε ο Ζαμαρή. Τι να πω, συμφωνώ απόλυτα φυσικά και πρέπει να σου πω, Ζαμαρία, ότι η στήριξη που μας προσφέρει είναι πολύτιμη, πολύτιμη για όλους εμάς. Και η στήριξη καθενός βουλευτή είναι πολύτιμη για όλους εμάς και βέβαια λόγω της δικής σου αξιοπιστίας αλλά και της ε, ισχύω που έχεις αν θέλεις, ε, την προβολή που έχεις ε, γενικώ, τη δημοτικότητά σου, όλα αυτά βοηθούν, είναι πολύτιμη συμβολή σου λοιπόν και γνωρίζουμε ότι θα, θα μας στηρίξεις. Όταν μιλάμε και λέμε ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να αναλάβει, φυσικά και υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό, μεταξύ άλλων ένας λόγος είναι ότι αυτό το project είναι ένα project που ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια και το οποίο όμως απέτυχε για 15 χρόνια αποτύχανε ακριβώς γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί σεφ στην κουζίνα ε, που μαγείρευαν ταυτόχρονα. Και ε, γι' αυτό τώρα νομίζω ότι κάπως ε, βελτιώνουμε προς αυτήν την κατεύθυνση και προχωράμε προς τα εμπρός. Αυτά που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει να ξέρεις και ότι η κυρία Λέα Σμιτ που είναι και διευθύντρια ε, του Μουσείου στη Βουδαπέστη που ανέφερες και είναι και μέλος ε, της διοίκησης μας βοηθά. Τα έχουμε όλα αυτά υπόψη μας. Προς την κυρία Τρούπελ θέλω να πω ότι φυσικά θα ήθελα να πω και να τονίσω ότι εκτιμήσαμε ιδιαίτερα την υποστήριξή σας σε πιο πολύπλοκες χρονικές στιγμές. Βέβαια ο καθένας μας δεν μιλάει μόνο ε, εκφράζοντα τη δική του προσωπική γνώμη, αλλά εκφράζοντα και την ε, άποψη τη δική του πολιτική ομάδα. Και η κυρία Τρούπερ δεν είχε πάντοτε εύκολο έργο όταν στήριζε το έργο αυτό. Θέλω να πω επίσης ότι φυσικά πρέπει, το είπε και ο κύριος Σταβάρης, ότι αυτό το μουσείο θα πρέπει, ναι με να το συσχετίσουμε, αν θέλετε να το συνδέσουμε με όλα τα μουσεία που υπάρχουν, αλλά όχι μόνο, να πάμε πολύ πιο πέρα. Το μουσείο μας πρέπει να έχει άμεση επαφή με τους οίκους της Ευρώπης, ε, τους οίκους του πολιτισμού, τα πανεπιστήμια, ε, τα μουσεία, αλλά και οποιαδήποτε, άλλη, οποιαδήποτε άλλο ίδρυμα ε, που έχει να κάνει με την κοινωνία των πολιτών και θα μπορούσε με τον ένα τον άλλο τρόπο να συμμετάσχει και να δώσει τις ιδέες του, όπως είπε ο φίλος Ταβάρης, για εκθέσεις προσωρινές, για παράδειγμα, διότι οι προσωρινές εκθέσεις νομίζω ότι θα διαδραματίσουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Επίσης θεωρώ ότι ακριβώς αυτό το πλαίσιο των προσωρινών εκθέσεων θα εκφραστεί η πολυφωνία, η πολυμορφία, κάτι που ενδεχομένως δεν θα το βλέπουμε τόσο πολύ στη μόνιμη έκθεση που θα είναι ένα αποτέλεσμα σύνθεσης. Στις προσωρινές εκθέσεις θα μπορούμε να εκφράσουμε την πολιτική πολυμορφία που χαρακτηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι και ο κύριος του έργου και παραμένει και θα εκφράζονται διαφορετικές σχολές σκέψης. Δεν ξέρω, κάποιοι μπορεί να πούνε ότι πρέπει να έχουμε μια έκθεση προσωρινή για τα δικαιώματα τη γυναίκα. Κάποιοι άλλοι μπορεί να μιλήσουν ότι θα πρέπει να έχουμε μια έκθεση για τον χριστιανισμό και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Μέσω λοιπόν αυτών των προσωρινών εκθέσεων θα μπορούμε να δείχνουμε ότι η κοινωνία μας παραμένει πολυπολιτισμική και πολυμορφη, και πλούσια. Α, για το προπολογισμό δεν μίλησα, ναι, ναι, ναι. Και για την κυρία Τρίπελ. Δεν μπόρεσε να ασχοληθεί το Προεδρείο με κάτι που δεν υπάρχει. Διότι υπάρχει πρόταση του Συμβουλίου, υπάρχει πρόταση του Συμβουλίου που κατά την άποψή μου δεν θα περάσει. Και αυτό, ε, τι να σας πω, θα ήταν επικίνδυνο το Προεδρείο να εκφραστεί για ένα παιδί το οποίο ακόμη δεν το έχουν συλλάβει γονείς του. Μπορεί ο πατέρας να έχει εκφράσει την πρόθεσή του, αλλά η μητέρα να μην είναι απόλυτα βέβαιη ακόμη. Λοιπόν, προς το παρόν, τα στοιχεία, τα οικονομικά που χειριζόμαστε στο πλαίσιο το, το δημοσιονομικό και τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα, είναι τόσο ταπεινά, αν μου επιτρέπετε, που κατά πάσα πιθανότητα δεν θα υπάρξει σημαντικός αντίκτυπος. Και το ίδιο ελπίζω να μην ισχύσει, να μην υπάρξει δηλαδή αντίκτυπος και στη δέσμευση της Κομισιόν να χρηματοδοτήσει τη λειτουργία του μουσείου. Γιατί και η λειτουργία του μουσείου, ε, πώς να το πω, θα είναι κάτι το έλασον ε, σε σχέση με τα συνολικά ποσά κατά που μιλάμε, αλλά και πάλι Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό δρόμο, καλό δρόμο. Να απαντήσω στον κύριο Ταβάρες για το 2014. 100 ε, χρόνια από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ε, ναι, όντως απασχολεί πολλές ε, ε κυβερνήσεις γιατί θέλουν πολλές να, τον επόμενο χρόνο να ασχοληθούν με το θέμα αυτό και στο Σεράγεβο, γιατί στο το Σεράγεβο είχαμε πει να είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα ε, για την Ευρώπη. Ε, το είχαμε προτείνει ως κοινοβούλιο, αλλά δεν ήταν για τεχνικούς λόγους ε, δυνατό. Έχουμε και τις γέφυρες για τον πολιτισμό και αυτό το πλαίσιο, το, αυτό το πρόγραμμα μάλλον θα περιλαμβάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Οπότε και εμείς, ανεξάρτητα από το νίκο της ιστορίας, που δεν είναι ακόμα έτοιμος, θα μπορέσουμε να ασχοληθούμε με, το, με τα 100 χρόνια από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε μπορούμε ίσως να συνδυάσουμε και τις δικές σας τις ε, ιδέες. Ωραία. Λοιπόν, δεν υπάρχουν άλλα ερωτήματα. Η κυρία Παλιαδέλη, όχι, εντάξει. Θέλετε μήπως εσείς να συμπληρώσετε κάτι, όχι, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε εδώ, κυρία Βαγκάλ, και σας εύχομαι καλή επιτυχία στη δουλειά σας. Είναι δύσκολη και να θυμίσω ότι το θέμα αυτό με το συμπόσιο ε, μας μας ενδιαφέρει πάρα πολύ πριν να είναι αυτός ο οίκος έτοιμος θα πρέπει όλοι οι εμπειρογνώμονε που, που ασχολούνται με αυτό να του αφήσουμε να ασχοληθούν με αυτό. Και όταν, αν, θέλουμε εμεί πάντα να κάνουμε το συμπόζιο την ίδιο καιρό και, θα, είναι και άλλοι 10 πάνω στο κεφάλι του και προσπαθούν να του πούνε πώ να κάνουν τη δουλειά του, δεν θα γίνει δουλειά. Α αφήσουμε του ανθρώπου να κάνουν τη δουλειά του, α αφήσουμε να, για να γίνει ο οίκο και μετά μπορούμε να σκεφτούμε να κάνουμε ένα συμπόσιο όπω το θέλουμε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη. Σημείο 5 Η συνάδελφος Κάμερα Εβερτ είναι η συγκήτρια, συνδεδεμένη τηλεόραση, έκθεση πρωτοβουλίας. Ε, ξέρετε ότι είναι πραγματικά πολύ δύσκολη, ήταν πολύ δύστοκη η γέννα αυτή της συνδεδεμένης τηλεόρασης. Πέτρα, έχεις το λόγο. Ja, vielen herzlichen Dank. Ευχαριστώ. Αν σκεφτείτε ότι αυτή η οδηγία για την οποία συζητούμε ε, μόλις πριν από τρία χρόνια μπήκε με την νέα μορφή της, ε, σε, τέθηκε σε ισχύ, τότε ε, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να συζητούμε σήμερα αυτό το θέμα και να μιλούμε πάλι για αναθεώρηση της οδηγίας μετά από τρία χρόνια. Μιλούμε λοιπόν για την συνδεδεμένη τηλεόραση. Έτσι, εκ πρώτη όψεω ε, φαινόταν σαν να μιλούσαμε μόνο για τεχνικά πράγματα, για τεχνικά θέματα, αλλά δεν ήταν έτσι. Γιατί στην ουσία μιλούμε για τη διαθεσιμότητα, για την προσβασιμότητα και την ειχνηλασιμότητα των ε, ε, προσφερόμενων τηλεοπτικών υπηρεσιών και είπαμε πότε θα γίνει αυτό, αν γίνει, εφόσον γίνει με ποια εργαλεία μπορεί να γίνει η σύγκληση και πώς μπορούμε να έχουμε μια ομοιόμορφη διαχείριση όλες αυτές της διαδικασίας. Ένα σημαντικό ε, τμήμα της συζήτησης είναι ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, είναι και πολιτιστικό αγαθό, αλλά είναι και ενημερωτικό αγαθό και γι' αυτό έχουν ιδιαίτερη σημασία στην ε, κοινωνία. Η ποικιλία λοιπόν των ΜΜΕ, η, ε, η ελευθερία της έκφρασης συμβάλλουν στην λειτουργία της δημοκρατικής μας κοινωνίας. Τα ΜΜΕ έχουν ρόλο και διασκεδαστή και ενημερωτικό ρόλο και πολιτιστικό. Ξέρουμε ότι χωρίς ε, νερό δεν μπορούμε να ζήσουμε και νομίζω ότι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τα ΜΜΕ ε, αποτελούν ένα ε, συνδετικό κρίκο για την κοινωνία μας. Για να μπορέσουμε λοιπόν να έχουμε τα ΜΜΕ αποτελεσματικά και αποδοτικά θα πρέπει να έχουμε με ένα συγκεκριμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα ΜΜΕ. Αυτός είναι ένας βασικός λόγος για τον οποίο εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στα κράτη-μέλη αποφασίσαμε την πολιτική για τα ΜΜΕ να μην την, ε, να μην την ε, αφήσουμε μόνο στα, ε, στην οικονομική πολιτική, αλλά να, τη θέσουμε σε ένα, να την θέσουμε σε ένα δικό της πλαίσιο, ακριβώς λόγω και του ιδιαίτερου χαρακτήρα της, των ΜΜΕ, αλλά και του ρόλου που έχουν να παίξουν στην κοινωνία. Και επίση είναι πεποίθησή μου ότι και η σύγκληση τη τεχνολογία που έχει να κάνει και με την υβριδική τηλεόραση δεν θα πρέπει να αλλάξει. Και νομίζω ότι οι τεχνικές εξελίξεις ε, θα μας ε, βοηθήσουν να προχωρήσουμε. Η υβριδική, ε, τα υβριδικά συστήματα λήψης είναι ένα σημαντικό μέσο, ένα σημαντικό βήμα για την σύγκληση. Υπάρχουν πάρα πολλές αριθμιστικέ αποφάσεις, τις οποίες έχουν, οι οποίες έχουν ληφθεί το προηγούμενο διάστημα. Στην οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα είχαμε αποφασίσει και δικαίως είχαμε αποφασίσει ότι οι γραμμικές υπηρεσίες ε, θα πρέπει να υπόκειται σε ένα συγκεκριμένο ε, πλαίσιο και οι μη ε, γραμμικές υπηρεσίε σε ένα λιγότερο αυστηρό πλαίσιο. Στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων είχα προσπαθήσει και εγώ να το παρουσιάσω αυτό για να, δείξω πώς ακριβώς θα λειτουργήσουν αυτά τα δύο διαφορετικά συστήματα για, τις δύο αυτές, για τα δύο αυτά είδη υπηρεσιών. Βεβαίω αυτέ οι υπηρεσίε έχουν διαφορετικέ επιπτώσει ε, στα, στα, στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουν την, ε, την κλασική γραμμική ε, προσφορά υπηρεσιών Και βεβαίω αυτό στα περισσότερα κράτη-μέλη διασφαλίζεται μέσω νομικού πλαισίου. Βεβαίω υπάρχει τεράστια, ε, είναι πάρα πολύ ελκυστική και η ψηφιακή τηλεόραση. Αν δούμε τα γραμμικά μέσα, Επειδή λοιπόν τα γραμμικά ε, μέσα θέλουμε να, είναι, να έχουν μεγαλύτερη απήχηση, πρέπει να έχουμε συγκεκριμένους κανόνες που θα τα διέπουν. Αυτή η διαφοροποίηση που είχαμε κάνει, που ε, αντικατοπτρίζεται και σε, αυτή την, ε, διαφορετική, σε αυτό το διαφορετικό επίπεδο πλαισίων που πλαισιώνουν αυτές ακριβώς τις υπηρεσίες, μπορεί να λύσει τα προβλήματα που δημιουργούνται κυρίως σε θέματα που μπορούν να, κυρίως σε μάλλον που μπορούν να λυθούν γρήγορα τα προβλήματα. Εμείς ως πολιτικοί δεν μπορούμε να είμαστε πάντα να παρακολουθούμε τις ε, ε, εξελίξεις, πρέπει να ε, μπορέσουμε να προπορευτούμε. Υπάρχει πρόσβαση και σε κλασικά βεβαίω ε, προγράμματα τηλεοπτικά, αλλά και στο ίντερνετ, κυρίω με αυτέ τι ε, νέε έξυπνε συσκευέ. Και πιστεύω ότι ε, σύντομα θα, γίνει, θα καταστεί δυνατή και η πλήρης σύγκληση. Η, μέσα από τις οθόνες θα μπορούμε στο μέλλον να έχουμε διάφορες υπηρεσίες, οι οποίε μέχρι τώρα υπόκεινται σε τελείω διαφορετικέ διαφορετικές οδηγίες. Μίλησα για τις ε, γραμμικές ε, οπτικοακουστικές υπηρεσίες, για τις μη γραμμικές. Έχουμε ε, υπηρεσίες που δεν καλύπτονται καν από την οδηγία, δεν έχουμε υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν καν στο πεδίο εφαρμογής οδηγίας. Υπάρχουν και ΜΜΕ τα οποία δεν υπόκειται σε καμία ευρωπαϊκή νομοθεσία. Μιλούμε για τα υβριδικά συστήματα λήψης πολύ συχνά για, μιλούμε για ε, υπηρεσίες που μπορεί κανείς να λάβει, υπηρεσίες ίντερνετ που μπορεί κανείς να λάβει μέσω της ε, οθόνης του. Επίσης, το περιεχόμενο, η προσφορά περιεχομένου είναι σημαντικό να, είναι, να υπόκειται σε πλήρη προσβασιμότητα και αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Όποιο ε, προσφέρει μια πύλη πληροφόρηση ή μια πλατφόρμα πάντα πρέπει να έχει μια επιλογή ε, για το ποια θα είναι τα περιεχόμενα που είναι διαθέσιμα και επίσης με ποιο τρόπο θα, υπάρξει προ... Ε, θα γίνει κάποια κατηγοριοποίηση, αν θα υπάρξουν προτεραιότητες και σε σχέση με την ε, τεχνολογία που θα τα καταστήσει όλα αυτά δυνατά. Τέλος, η ο πάροχος της πλατφόρμας ή της πύλης ή ο κατασκευαστής ακόμα των συσκευών μπορεί να ελέγξει και βεβαίω αυτά τα τρία μπορεί να είναι είτε μια εταιρεία είτε ένα άνθρωπο. Μπορεί να ελέγχει λοιπόν την ε, πρόσβαση ε, στο σχετικό περιεχόμενο και έτσι η πάροχοι των πλατφορμών, οι, οι, ε, οι κατασκευαστές των συσκευών μπορούν να έχουν το ρόλο ενός gatekeeper. Νομίζω λοιπόν ότι θα είναι απαραίτητο, κυρίως για τούτη την οδηγία, αυτά τα νέα δεδομένα να μπορέσουμε να τα ενσωματώσουμε. Γιατί αλλιώς μπορεί να διακυβεύσουμε την ελευθερία της προσφοράς περιεχόμενου και η βασική θέση που έχουν οι πάροχοι των πλατφορμών μπορεί να είναι βλαβερή για τις υπηρεσίες τις υβριδικές ακριβώς γιατί είναι πολύ συγκεκριμένες οι ε, προϋποθέσεις ε, σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να προκύψει μια νέα πλατφόρμα ενημέρωσης. Βεβαίως πρέπει να διασφαλίσουμε τον ε, δίκαιο ανταγωνισμό, για τον οποίο μονίμως μιλούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίκαιο ανταγωνισμό λοιπόν μεταξύ των, της προσφοράς, επί τη βάση όμως ενιαίων προϋποθέσεων ανταγωνισμού ενιαίων, τεχνολογικώς ενιαίων, ανοιχτό, ανοιχτών και ε, ε, διαλειτουργικών συστημάτων που θα προσανατολίζονται προς την αγορά και για τους παρόχους αλλά και για ε, την, τον τελικό χρήστη. Επίσης, η χνηλασιμότητα και η προσβασιμότητα της παροχής γίνεται κεντρικό θέμα της εξασφάλισης της ε, πολυμορφίας των υπηρεσιών αυτών και η πρότασή μου είναι ότι τα μέχρι τώρα συστήματα της προηγούμενη ε, οδηγία θα πρέπει να εξελιχθούν γιατί θεωρούμε ότι μόνο λίγα είναι αυτά τα οποία έχουν τους, τους ε, πόρους ώστε να μπορέσουν να έχουν ε, επιρροή. Οι πόροι όμως αυτοί πάντα χρησιμοποιούνται από τις κλασικές υπηρεσίες. Η ψηφιοποίηση επίσης του περιεχομένου είναι πολύ σημαντικό θέμα και Βεβαίω, ανεξάρτητα από, το, από τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτό, πρέπει, πρέπει να είναι ε, τα, τα περιεχόμενα αυτά ψηφιοποιημένα και διαθέσιμα για όλους. Βεβαίω, τώρα αυτό θα πρέπει να το δούμε σε σχέση και με το με ποιο τρόπο θα γίνει. γιατί κανεί ε, μπορεί να μην ξέρει καν αν λαμβάνει ένα σήμα γραμμικό ή αν είναι ψηφιακό ή αν είναι δορυφορικό ή μέσω ποιου, τι ακριβώς καταναλώνει και μέσω ποιου καναλιού. Πρέπει λοιπόν ε, να αναγνωρίσουμε ότι αυτή ακριβώς η ε, σπάνιδα των πόρων επηρεάζει και την, και την προσβασιμότητα και την κλεινασιμότητα του σήματος μέχρι τώρα Δικαίω είχαμε ρυθμίσεις must carry. Νομίζω ότι στο μέλλον όμως η τεχνική ακριβώς και η εξέλιξη, θα πρέπει να, η εξέλιξη τεχνολογίας θα πρέπει να συμπληρωθεί και με τους must be found κανόνες, υποχρεώσει δηλαδή της ανείχνευσης. Ακριβώς αυτές ε, οι υβριδικές πλατφόρμες θα πρέπει να είναι εύκολα ανοιχνεύσιμες και τα κράτη-μέλη θα πρέπει είτε μέσω δημοσίων ε, συμβάσεων να το πράξουν, είτε αυτοί που θέλουν ε, να ε, χρηματοδοτήσουν κάποιοι ιδιώτες, ας πούμε, θα μπορούσαν να το αναλάβουν. Ή ακόμα και άνθρωποι που θέλουν να εξασφαλίσουν την ποιότητα της, του πλουραλισμού στα ΜΜΕ. Μιλάω δηλαδή και για αυτορύθμιση. ή έτσι όπως το λέμε εμείς στη Γερμανία η ρυθμισμένη αυτορύθμιση. Ένα τέτοιο σύστημα μάλλον στο μέλλον θα πρέπει να λάβει πολύ σημαντικό ρόλο. Όποιος λοιπόν θα υπόκειται σε αυτούς τους ε, αυστηρούς κανόνες ε, της οδηγίας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να έχει μια δεσπόζουσα θέση σε μια πλατφόρμα και νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά ποιε είναι αυτέ οι ε, νέε μορφέ ε, ε, κινήτρων που θα μπορούσαμε να θέσουμε για, την, για να μπορέσει κανεί να, να αποφασίσει κανεί να υποστεί όλου αυτού του αυστηρού κανόνε τη αυτορύθμιση. Επίση, οι κατασκευαστέ των συσκευών αλλά και οι πάροχοι του περιεχομένου αυτού θα επηρεαστούν πολύ. και βεβαίω θα πρέπει να μην δημιουργήσουμε για κάποιου δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Να μην δημιουργήσουμε δηλαδή μονοπόλια σε μία ε, πλατφόρμα. πούμε κάποιο μπορεί να βάλει πολλά λεφτά και να ε, πάρει ουσιαστικά να αγοράσει την, την πλειοψηφία του μεριδίου της αγοράς. Αυτό θα πρέπει να το αποτρέψουμε μέσω συγκεκριμένων κανόνων. Νομίζω ότι στα πλαίσια και των τεχνικών ε, αλλαγών και εξελίξεων θα πρέπει να θέσουμε κάποια ερωτήματα και να ξανασκεφτούμε κάποια πράγματα. Για του ε, παρόχου ε, γραμμικών υπηρεσιών, σε ό,τι αφορά τι διαφημίσει, έχουμε θέσει πολύ συγκεκριμένου κανόνε. Και αυτό ήταν ε, πολύ καλό, το είχαμε μελετήσει, αλλά αν μιλούμε για ακόμα πιο ε, μεγάλη σύγκληση σε ό,τι αφορά την τεχνική, και να λάβουμε υπόψη ότι οι, οι διαφημίσεις θα είναι ανεξάρτητες στο μέλλον από τους γραμμικούς παρόχους ή τους μη γραμμικούς παρόχους. Και σύμφωνα με τους τρέχοντες κανόνες, οι πάροχοι μη γραμμικών υπηρεσιών και οι πάροχοι υπηρεσιών που δεν περιλαμβάνονται στην οδηγία που δεν υπόκειται δηλαδή σε κανένα κανόνα, είναι, βρίσκονται στον ίδιο ανταγωνισμό με τους, ε, γραμμικούς, με τους παρόχους γραμμικών υπηρεσιών και μπορούν να στείλουν το δικό τους σήμα ε, ή το, δικό τους περιεχόμενο. Αυτό ουσιαστικά οδηγεί σε στρέβλωση του ανταγωνισμού, γιατί έτσι ο ιδιώτης πάροχος προφανώς ε, βρίσκεται, δεν έχει το πλεονέκτημα που έχει ο γραμμικός πάροχος και ο οποίος δεν υπόκειται σε, καμία, σε κανέναν κανονισμό για τις διαφημίσεις. Οπότε, στο κείμενό μου λέω ότι πρέπει να μελετήσουμε τι θα γίνει με την ευελιξία ή την απελευθέρωση αυτών των κανόνων για τις ε, διαφημίσεις. Δεν μιλάω για το ότι θα πρέπει να πούμε οι διαφημίσεις θα πρέπει να, να μην υπόκειται σε κανέναν σε κανένα κανόνα. Όχι, δεν λέω καθόλου αυτό. Αλλά αυτό που λέω είναι να θέσουμε το ερώτημα. Χρειάζεται αυτό ο κανόνα των συγκεκριμένων λεπτών διαφήμιση που πρέπει να υπάρχουν στι διάφορε εκπομπέ, ή μήπω θα πρέπει να μιλήσουμε για μια ημερήσια, α πούμε, καταποκοπή χρονική περίοδο διαφημίσεων. Ίσως αυτό να οδηγήσει σε πιο υψηλή ποιότητα προγράμματα. Αν, α πούμε, αποφασίσει κάποιο, έχω ένα πολύ ωραίο παιδικό πρόγραμμα, δεν θα το επιβαρύνω με διαφημίσει, αλλά έχω τη δυνατότητα σε, ένα άλλο, σε μια άλλη εκπομπή, σε ένα σοου ή σε μια ε, εκπομπή ε, ενημερωτική, να βάλω τις, ε, να βάλω τις διαφημίσεις μου εκεί. Αυτό ίσως θα μπορούσαμε να το αφήσουμε λοιπόν στην αγορά να το αποφασίσει αν δούνε οι αγορέ ότι οι καταναλωτέ φεύγουν ε, μαζικά από τα προγράμματα του και δεν τα παρακολουθούν ή κλείνουν την τηλεόραση, τότε όντω μπορεί και αυτοί να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης τους. Επίσης, μιλούμε για πλουραλισμό στα ΜΜΕ και λέμε ότι αυτή την, ε, αυτόν τον πλουραλισμό θέλουμε να τον διατηρήσουμε και έχουμε πάρα πολύ καλές ε, ε εκθέσεις και από τον Ιβο Μπέλετ για τα, ραδιοφωνικά, ε, για σήματα, αλλά αν θέλουμε να έχουμε ένα τέτοιο σύστημα και δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τότε θα πρέπει και στους ιδιώτες παρόχους να δώσουμε την δυνατότητα να, ε, κερδίσουν αυτά τα χρήματα που τους χρειάζονται για να μπορέσουν να παρέχουν ποιοτικά προγράμματα. Γι' αυτό σας ζητώ ακριβώς για τον κανονισμό για τις, ε, ε, για τις διαφημίσεις, να μην τον καταργήσουμε τελείως, αλλά να μιλήσουμε για μια έτσι, ευελιξία ή απελευθέρωση αυτού του κανόνα. Και να δούμε Πώ θα μπορέσουμε να μην, δημιουργήσουμε στρέβλωση του ανταγωνισμού που μπορεί βεβαίω να βλάψει και την, τον πλουραλισμό των ΜΜΕ. Επίση, αυτή η οδηγία θα πρέπει να ε, διαφοροποιηθεί, θα πρέπει να εξελιχθεί μάλλον σε ένα ακόμη σημείο, στα υβριδικά, στις υβριδικές, στα υβριδικά συστήματα παροχή. Γιατί οι, α, κατασκευαστές ε, των συσκευών στο μέλλον θα έχουν τελείω διαφορετική θέση από αυτή που ξέραμε μέχρι τώρα. Επίση, σημαντικό θα είναι και η, ο πλουραλισμό και στην προσφορά αλλά και, στις, και στην άποψη. Οπότε εδώ θα πρέπει να έχουμε αυστηρούς κανόνες. Επίσης, οι συσκευέ, οι πλατφόρμες και οι πύλες θα πρέπει να βασίζονται σε μια ανοιχτή, σε ένα ανοιχτό και διαλειτουργικό πρότυπο, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε θέματα διακριτικής μεταχείρισης και ουδετερότητας στην πρόσβαση. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι το σημείο της ανάμειξης προγραμμάτων, που θα πρέπει να παραμείνει απαράλλαχτο κάποιο που στέλνει την εκπομπή του οποιοδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο και τον κάνει, πρέπει να είναι σίγουρο ότι δεν θα, δεν θα συγχωνευτεί με άλλο περιεχόμενο που προσφέρει άλλο πάροχο. Επίσης, αν δεν ε, υπάρχει έγκριση από τους ε, από τους παρόχους ή αν δεν υπάρχει έγκριση από τους, ε, από τους καταναλωτές ε, κάποιες ε, εκπομπές θα πρέπει να καταργηθούν πλήρως. Επίσης, η ιδιωτικότητα που θα μπορεί να διασφαλίζεται μέσω της συσκευές κυρίως όταν μιλούμε για πολύ στάνταρ συσκευές. Και αυτό βεβαίω θα πρέπει να το ε, συνδυάσουμε και με την αναλογικότητα και με την αποθήκευση των δεδομένων, αλλά και με την πλήρη διαφάνεια στη μεταβίβαση δεδομένων και για την χρήση και για την περαιτέρω διαβίβαση δεδομένων. Και πρέπει βεβαίω να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα, γιατί συνήθω μιλούμε για τέτοια συστήματα, μόνο, θα μπορούν να ε, συλλέγονται μόνο με την έγκριση, με τη συγκατάθεση του καταναλωτή. Έτσι ώστε να διευκολυνθεί η παροχή μιας υπηρεσίας. Τελευταίο σημείο. Η χρήση ανωνύμως των ΜΜΕ η ανώνυμη χρήση θα πρέπει και στο μέλλον να υπόκειται σε κανόνες, θα πρέπει να γίνει ένας, έτσι, μια αξιολόγηση των, του προφίλ των χρηστών, της χρήσης των χρηστών, ίσως να κάνουμε και μια ανάλυση των, των, των διευθύνσεων του πρωτοκόλου που χρησιμοποιούν οι χρήστες και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το εξασφαλίσουμε και νομικώς. Ε, είτε γίνει αυτό μέσω της οδηγίας είτε μέσω κάποιου άλλου νομοθετικού κειμένου. Αυτά είναι, αυτές είναι οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεσή μου. Θα δείτε ότι στο ένα ε, ή στο άλλο σημείο ήμουν αρκετά αυστηρή, ε, είναι αρκετά σύντομη η έκθεση γιατί πάντα έχω έτσι ένα φόβο με τους χαρακτήρες που μου διατίθενται όταν μιλούμε για εκθέσεις πρωτοβουλίας. Ίσως θα, μπορούσαμε σε κάποια, θα μπορούσα σε κάποια σημεία να είμαι λίγο πιο γλαφυρή, αλλά προσβλέπω στα δικά σας σχόλια. Θα ήθελα να σας καλέσω επίσης στις 16 Μαρτίου εδώ στο Κοινοβούλιο θα κάνω μία μικρή παρουσίαση ε, με, το, με τη βοήθεια του Ινστιτούτου για την, ε, ραδιοφωνική, ραδιοφωνική τεχνολογία ε, από το Μόναχο ε, για να δείξουμε πώς ακριβώς λειτουργεί αυτή η υβριδική παροχή, η υβριδική υπηρεσία. Ε, ε, πώς λειτουργούν τα ευρυδικά συστήματα λήψη, πώ λειτουργούν οι ευρυδικές τηλεόρασει, Όποιο έχει χρόνο, 16 Μαρτίου είναι ευπρόσδεκτος. Έτσι ώστε για να δείτε και ζωντανά τι ακριβώς σημαίνει η ευρυδική τηλεόραση και ελπίζω ότι οι ε, περαιτέρω συζητήσει μας θα εμπλουτιστούν μόλις έχουμε και αυτή την ευκαιρία να δούμε από κοινού αυτή την παρουσίαση. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ Πέτρα. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σου. Η Κομισιόν είχε πει ότι θα κάνει μια πράσινη βίβλο, νομίζω τον Απρίλιο είπε θα την, θα την δημοσιεύσει. Ίσως να μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτά που είπες εσύ. Έχω τέσσερις συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο. Η κυρία Φεράν και μετά η κυρία Τρούπελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχάς την Πέτρα. Νομίζω ότι στην έκθεση πρωτοβουλία της Είναι πραγματικά πλήρης η παρουσίαση της κατάστασης και τα ερωτήματα επίσης για την περαιτέρω εξέλιξη της ε, ε, τεχνολογίας ε, περιλαμβάνουν όλες τις δυνατές υπηρεσίες, όχι μόνο τη συνδεδεμένη τηλεόραση, γιατί μιλούμε και για το ίδιο πρόβλημα και για άλλους για, άλλα είδη συσκευών, ας πούμε το είναι ταμπλέτα μου όταν εγώ θέλω να δω τηλεόραση μέσω της ταμπλέτας μου κτλ. πρόβλημα λοιπόν, το πρόβλημα δεν, είναι, δεν έχει να κάνει μόνο με την ε, συνδεδεμένη τηλεόραση, αλλά και με όλες τις έξυπνες συσκευέ που ε, παρέχουν τέτοιου είδου υπηρεσίες. Ε, θεωρώ ότι είναι πολύ καλή έκθεση της Πέτρα. Μας δίνει μια πολύ καλή γενική εικόνα για, την, ε, για τα θέματα που, που αφορούν και την πολιτική ΜΜΕ και νομίζω ότι είναι σημαντικό να σκεφτούμε οι κανόνες που ίσχυαν μέχρι τώρα πώς μπορούν να, ε, να στοχοθετηθούν καλύτερα σε ό,τι αφορά τι ομάδε στόχου, δηλαδή του παρόχους γραμμικών υπηρεσιών, μη γραμμικών υπηρεσιών κτλ. Σε έναν ε, κόσμο που συγχωνεύονται τα πάντα, νομίζω ότι θα πρέπει να ξανασκεφτούμε πολλά πράγματα που μέχρι τώρα τα θεωρούσαμε ως ε, δεδομένα. Θα πρέπει όντως να έχουμε συγκεκριμένους κανόνες που πρέπει βεβαίως να δομηθούν διαφορετικά σε σχέση με τα όσα υπάρχουν τώρα στην οδηγία. Το θέμα της, ε, ε, της εξειδίκευσης για το ραδιόφωνο ίσως να είναι λίγο πιο δύσκολο να λυθεί γιατί υπάρχουν πολύ περισσότερες προσφορές, υπάρχει νέα τεχνολογία, υπάρχουν ουδέτερες ε, λύσεις που χρειάζονται. Ας πούμε, σε ό,τι αφορά τη διαφήμιση και τις προστασίες των παιδιών, των νέων, θα μπορούσαμε να έχουμε ε, μια ουδέτερη τεχνολογία και σε ό,τι αφορά την ε, ισότητα των όπλων για όλους, αλλά ίσως θα μπορούσαμε για κάποιο συγκεκριμένο περιεχόμενο να παραμείνει έτσι μια διαβαθμισμένη ε, δυνατότητα προστασίας. Όταν δηλαδή θέλουμε να έχουμε προστασία για τα παιδιά στο διαδίκτυο, θα πρέπει να έχουμε πιο υψηλούς, πιο αυστηρούς κανόνες για την προστασία τους. Οπότε ας υπάρχει μια ευελιξία έτσι ώστε και στο μέλλον να μπορούμε να διευκολύνουμε και την περαιτέρω, και την περαιτέρω χρηματοδότηση αυτής της παροχής των υπηρεσιών. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να, δούμε, να βρούμε νέες λύσεις για το πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε μια πιο λογική κατάσταση. Επίσης, το μέλλον, το δημόσιο και το ιδιωτικό, ε, τα, τις δημόσιες και τις ιδιωτικές υπηρεσίες, παροχές υπηρεσίας, πώς μπορούμε να τις ρυθμίσουμε για να εξασφαλίσουμε, και για μένα αυτό είναι σημαντικό, ότι για κάποιους τομείς θα πρέπει να μπορούμε να εγγυηθούμε την ε, ε, ελευθερία της διαφήμισης. Ας πούμε, σε ενημερωτικές εκπομπές κτλ αυτό είναι ένα κομμάτι της, ε, το, της δημοκρατίας μας. Παράλληλα με αυτό θέλουμε να έχουμε ανέλεγκτες, ανεξέλεγκτες διαφημίσεις ή θέλουμε να λαμβάνουμε τις πληροφορίες που μπορούν να προκύψουν και μέσω της συνδεδεμένης τηλεόρασης. Πρέπει να βρούμε λύσεις, πρέπει να βρούμε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα πέρα από, την ε, νομοθετική, από τον νομοθετικό διαχωρισμό του, των γραμμικών και των μη γραμμικών υπηρεσιών, θα πρέπει αυτό τον ε, ε, διαχωρισμό να τον κάνουμε για, τα, για τους καταναλωτές, γιατί προς το παρόν δεν φαίνεται. Η Πέτρα το είπε σαφώς, ότι όντως κάποια στιγμή δεν θα μας λαμβάνουν στο σοβαρά υπόψη τους. Εγώ έχω ένα γραμμικό πρόγραμμα, είμαι σε μια μη γραμμική υπηρεσία, έχω το βίντεο που τρέχει, μπαίνω σε ένα δωμάτιο και βλέπω ε, ένα συνδεδεμένο μέσο, δεν θα ξέρω αν όντω αυτό είναι συνδεδεμένο ή όχι. Δεν είναι πια διαφανεί οι κανόνε, τουλάχιστον για μένα ω καταναλωτή. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα με κίνητρα, όπω είπε και η Πέτρα. Είναι σκόπιμο. Και θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση για το πώς θα είναι αυτό το, το σύστημα των κινήτρων. Ίσως να μπορούσαμε να μιλήσουμε για ένα σύστημα αδειοδότηση με συγκεκριμένα κριτήρια, κάτω από, δηλαδή από ποιες προϋποθέσεις ένα ειδικό ε, περιεχόμενο μπορεί να λάβει και ειδικού ε, κανόνες για την προβολή του. Ίσως αυτό θα μπορούσε να, το, να μπει στην έκθεση. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά ακόμη που θα πρέπει βεβαίως να τα δούμε και σε ό,τι αφορά το ε, νομοθετικό κείμενο και υπάρχουν και ερωτηματικά τα οποία επίση πρέπει να θέσουμε για το πώ μπορούν οι τεχνικοί και πώ μπορούμε να δομήσουμε αυτού του τεχνικού και του ε, νομοθετικού κανόνε. Είχαμε κανόνε, κανονισμού, οδηγίε για την, ε, για την τηλεόραση, για τι τηλεπικοινωνίε. είχαμε κανόνε για, ε, για την προσία των νέων. Πώ μπορούμε όλα αυτά να τα ενοποιήσουμε για ένα μέσο που θα συγχωνεύει, που θα συνδυάζει τελικά τα πάντα. Νομίζω ότι και σε άλλες επιτροπές, όχι μόνο εδώ, θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό και με την online προσφορά, με τις προσφορές στις έξυπνες συσκευέ. Για να δούμε πώς θα τα συνδυάσουμε. Μιλούμε για έναν ε, κόσμο που συνδέεται όλο και περισσότερο. Οι πλατφόρμες επίσης είναι πολύ σημαντικές. Η προσβασιμότητα είναι σημαντική, η ουδετερότητα είναι επίσης σημαντική και πρέπει να είναι εγγυημένη. Η χνηλασιμότητα επίση είναι πολύ σημαντικό σημείο και η Πέτρα το είπε. Θα πρέπει να προσέξουμε ώστε οι παροχοί των, των πλατφορμών ή οι κατασκευαστές των διαφόρων συσκευών να μην θεωρήσουν τους εαυτούς τους ως, κύριο, ως κύριοι του, της πληροφόρησης. Έχουμε και τους κανόνες ε, must carry, έχουμε και τους ε, κανόνες ε, must be found. βεβαίως πρέπει να παραμείνει ο πλουραλισμός των μέσων. Και επίσης σημαντικό είναι σε ό,τι αφορά τη διαλειτουργικότητα να βρούμε δυνατότητες έτσι ώστε τα τεχνικά πρότυπα να μην μας οδηγήσουν στο να βρίσκουμε κάποιο περιεχόμενο μόνο στη μία πλατφόρμα και όχι στην άλλη. Επίση, η ευθύνη των κατασκευαστών ως gatekeepers είναι πολύ σημαντική. Το ερώτημα είναι ποια ευθύνη υπάρχει απέναντι τώρα στην προστασία των νέων, ε, κυρίως σε έναν πάροχο πλατφόρμας. Ας πούμε το μεσημέρι είναι ε, παραδοσιακά αφιερωμένες οι ώρες αυτές σε παιδικές ε, εκπομπές. Πώς μπορούμε λοιπόν όταν, ε, να είμαστε σίγουροι ότι όταν εγώ αφήνω το παιδί μου να δει ένα παιδικό στην τηλεόραση, πώς θα είμαι σίγουρη ότι δεν θα προκύψει, δεν θα βγει στην τηλεόραση κάτι άλλο που δεν θέλω να δει το παιδί μου. Αυτό πρέπει να δούμε πώ μπορούμε να το κάνουμε μέσω των παρόχων των πλατφορμών. Ή εν πάση πρέπει να θέσουμε τα ερωτήματα αυτά και να τα συζητήσουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να... δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε μια ευέλικτη δυνατότητα σε ό,τι αφορά την... Ε, τις διαφημίσεις. Είπαμε για, ε, για τα ε, παιδικά προγράμματα και για τις ενημερωτικές εκπομπές και τις ειδήσει, αλλά να μην έχουμε αυτό τον αυστηρό κανόνα όπως είχαμε στο παρελθόν με τα 12 λεπτά, γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί να διατηρηθεί. Χρειάζεται ευελιξία στο σύστημα, πρέπει να δημιουργηθεί ένα επίπεδο όπου στις διάφορες προσφορές υπηρεσιών θα μπορεί να υπάρξει και ένα λογικό πλαίσιο ανταγωνισμού. Πάντα είναι δύσκολο τέτοια θέματα μεγάλα να τα συμπεριλάβει κανείς και να τα καλύψει πλήρως σε μια έκθεση. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι όταν κανείς έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων για να περιγράψει όλα αυτά τα θέματα και ελπίζω ότι θα είναι καλή η συνεργασία μας και μέσω κάποιων ε, τροπολογιών ε, θέλω να πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε ένα πάρα πολύ καλό κείμενο. Ούτως ή άλλως το κείμενο της ε, Πέτρας είναι πολύ καλό. Γιατί νομίζω ότι όντω είναι ένα θέμα το οποίο δεν αφορά μόνο τι ε, τεχνικέ επιτροπέ. Μιλούμε για περιεχόμενο, μιλούμε για τη διαβίβαση περιεχομένου, μιλούμε για ε, δημοκρατικέ δομέ, μιλούμε για ενημέρωση, για πολιτισμό και αυτό θα πρέπει να καταστεί σαφέ. Δεν μιλούμε μόνο για τεχνολογία. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Τρίπελ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Πέτρα για την ε, πολύ καλή παρουσίαση που έκανε και για, την, ε, για, το, για το, την τροφή για σκέψη που μας έδωσε. Να πω κι εγώ δύο πράγματα. Τα είπες και εσύ βέβαια Πέτρα και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά και για την ε, πολιτική στοχοθέτηση αυτής της έκθεσης. Καταρχάς είπες ότι όλοι μαζί θα πρέπει ε, παρόλο που μπορεί να έχουμε δουλέψει πολύ ε, πάνω σε αυτή την ε, ε, οδηγία, ότι μας έχει προσπεράσει η τεχνολογία, η ψηφιακή τεχνολογία. Όντως, τα πράγματα, οι τεχνολογικές εξελίξεις κινούνται τόσο γρήγορα που πάντα είναι δύσκολο να βρούμε τις, τις απαντήσεις. Πάντα βρισκόμαστε ένα βήμα πιο πίσω και αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι είναι σωστό και αυτή είναι και η πολιτική μας ευθύνη να μιλούμε για μια ε, σωστή ε, ρύθμιση. Βεβαίως ε, είναι σωστό αυτό που λες και το συμμερίζομαι κι εγώ. Και επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι πρέπει να ξεκαθαριστεί για την, για την προσφορά των ΜΜΕ ότι μιλούμε για τον διπλό χαρακτήρα των ΜΜΕ είναι και προϊόν αλλά είναι και πολιτιστικό αγαθό και όντω πρέπει να ρυθμιστεί διαφορετικά σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα αγαθά τη αγορά. Γι' αυτό αυτή η οδηγία δεν μπορεί να μιλά μόνο για την οικονομική πτυχή και για τον ανταγωνισμό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό σημείο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλε πολιτικέ δυνάμει βέβαια που έχουν άλλε απαιτήσει. Είναι λοιπόν σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, μια που μιλούμε και για τη σύμβαση της UNESCO για την ε, προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς η οποία επίσης έχει κωδικοποιηθεί. Επίσης, πρέπει να καταλάβουμε, όπω το είπε και η Ζαμπίνε, ότι οι κατασκευαστές των συσκευών δεν θα είναι οι κύριοι της ε, πληροφορίας και ότι μιλούμε για gatekeepers. Και βεβαίω, εφόσον πρόκειται για gatekeepers, πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι οι κανόνε που θα του διέπουν. Γιατί είναι σαφέ ότι οι πιο ισχυροί οικονομικά κύκλοι και οι πιο ε, εξοικειωμένοι με το, με το πολύ γρήγορα ε, περιεχόμενο και τις μεγάλες ε, αλλαγέ προφανώ μπορούν να χρησιμοποιήσουν την θέση του. Πρέπει λοιπόν να υπόκειται και αυτοί σε συγκεκριμένου κανόνε. Τη βασική λοιπόν προσέγγιση είναι, τη βρίσκω σωστή γιατί ότι θα πρέπει δηλαδή να είναι σωστή η ρύθμιση που θα βρούμε. Επίσης, κάτι άλλο που είπε η Πέτρα και είναι σημαντικό, είπε ότι δεν έχουμε την, για, τη διανομή του περιεχομένου, έχουμε μια κατηγορία σπάνιδας στο, για το περιεχόμενο αυτό, για το πού καταχωρούνται αυτά τα περιεχόμενα. Και από τη συζήτηση βλέπουμε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Το θέμα είναι το θέμα πια δεν είναι από πού ε, υπάρχει αυτή η, πού, πού υπάρχει αυτή η σπάνιδα, αλλά πού ακριβώς ε, μπορούν να καταχωρούνται όλα αυτά τα περιεχόμενα. Αυτό είναι σημαντικό γιατί ξέρουμε ότι στον ψηφιακό, ο ψηφιακός κόσμος είναι ένα πάρα πολύ καυτό θέμα και υπάρχουν πολλοί που υπαρχει αυτη η που υπαρχει αυτη η σπανιδα αλλα που ακριβως μπορουν να καταχωρουνται ότι κοσμος ε, ειναι ενα παρα πολυ καυτο θεμα και υπαρχουν πολλοι που λενε οτι δεν υπάρχει καμία σπάνιδα πια και νομίζω ότι αυτό που λες εσύ το έκανε πραγματικά πολύ παραστατικό γιατί πραγματικά πρέπει να αφοσιωθούμε σε αυτό το πρόβλημα και πρέπει να καταλάβουμε πού ακριβώς υπάρχει η έλλειψη και προς τα πού έχει μεταφερθεί το πρόβλημα αυτό. Τώρα, για τη ρύθμιση για τις διαφημίσεις. Ναι, όντως υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει δυνατότητα να καταλήξουμε σε στρέβλωση του ανταγωνισμού ακριβώς γιατί οι γραμμικές ε, υπηρεσίε ε, ρυθμίζονται πολύ πιο αυστηρά από άλλες. Ευελιξία λοιπόν, ευελιξία και στα ποσοτικά δεδομένα. Και επίσης να μιλούμε και για ποιοτική ρύθμιση. Εμείς ε, εδώ θυμόμαστε τη συζήτηση που είχαμε κάνει για, για το δίκτυο και για την ανταλλαγή, τη μη εμπορική και την εμπορική. Το να το ορίσουμε αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο και για να γίνει αυτό έπρεπε να οριστούν οι κανόνες για τις, ε, για τις Υπάρχουν ε, κανόνες που δεν ήταν ε, διαφανείς. Χρειαζόμαστε λοιπόν μία πολιτική συζήτηση για το πώς θα λύσουμε το θέμα της ε, διαφήμισης στις διάφορες πλατφόρμες. Αν, αν δεν υπάρχουν να το συζητήσουμε, αν θέλουμε να υπάρχουν, κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα υπάρχουν διαφημίσεις. Συμμερίζομαι επίσης αυτό που λέει η Πέτρα για το ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει ε, συγχώνευση ή ανάμειξη των διαφόρων περιεχομένων και αυτό πρέπει να γίνει μέσω νομικών κανόνων. Και ένα τελευταίο σημείο, σημαντικό για την πολιτική μας συζήτηση και γι' αυτό θέλω να το πω, το θέμα της πιστοποίησης. Λέμε ότι υπάρχει, υπάρχουν κάποια ε, πρότυπα τα οποία πρέπει να είναι καλύτερα και πρέπει να φαίνονται περισσότερο από άλλα. Υπάρχει δηλαδή ένα σύστημα ρύθμιση για το πώ καταλήγει κανεί αυτή την πιστοποίηση. Έχει οριστεί αυτό πολιτικά. Τι θέλουμε δηλαδή για την προστασία των νέων στα μέσα, τι θέλουμε για του άλλου τομεί και μετά πρέπει και οι, προ... και οι πάροχοι να προσπαθήσουν να πάρουν αυτή την πιστοποίηση έτσι ώστε να έχουν καλύτερη θέση στην καταχώρηση. Αυτό γενικώ είναι πολύ λογικό. Μπορούμε να το συνεχίσουμε να το συζητούμε αλλά νομίζω ότι αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτό, ότι συνδέοντας την γραμμική προσφορά και την ε, προσφορά μέσω διαδικτύου υπάρχουν κάποια πρότυπα τα οποία ζητά η κοινωνία και δίνει και ε, περισσότερα, έτσι, περισσότερους ε, πόντους σε όσους έχουν αυτή την επιστοποίηση. Πρέπει να υπάρχει η ελευθερία την οποία όμως πρέπει να κατανοούμε σωστά. Αυτά και ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Χίρσου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και από μένα, ευχαριστώ την Πέτρα για την ε, έκθεση. Περιλαμβάνει κάποια σημεία τα οποία βεβαίως υποστηρίζουμε και φυσικά θέλουμε να, τα να τα συζητούμε μπορούμε να συζητήσουμε και φιλοσοφικά και επιστημονικά, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας πάντα το τι θέλει ο καταναλωτής. Και νομίζω ότι καλό θα ήταν να, να, ξέρουμε ότι ο καταναλωτής είναι αυτός που ανάβει την τηλεόραση και αυτός που, αυτό που βλέπει μπορεί να είναι από το ίντερνετ, μπορεί να είναι από γραμμική παροχή, από μη γραμμική, αλλά κανένας δεν πρόκειται να κάτσει να σκεφτεί από πού έρχεται αυτή η εκπομπή που βλέπω, από ποιο είδος παροχής. Πρέπει επίσης να σκεφτούμε Μάλλον υπάρχουν δύο τρόποι να λύσουμε το πρόβλημα. Είτε θα προσπαθήσουμε αυτή την προσφορά της μη γραμμικής παροχής, δηλαδή μέσω διαδικτύου κτλ, να την, να την ε, θέσουμε μέσα στο πλαίσιο των κανόνων που έχουμε τώρα. Και αν, κάνουμε, αν ακολουθήσουμε αυτή την άγουσα θα πρέπει να ελέγξουμε βεβαίως, θα πρέπει να υπάρξει έλεγχος και εποπτεία και πρέπει να πω ότι δεν νομίζω ότι το ίντερνετ μπορούμε με κάποιο τρόπο να το υποπτεύσουμε και επίσης δεν θέλουμε και να το υποπτεύσουμε. Οπότε αυτός ο δρόμος νομίζω δεν είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Άρα πρέπει να ακολουθήσουμε τη δεύτερη εναλλακτική και να πούμε στους καταναλωτές, αγαπητέ καταναλωτή, αν ανοίξει σήμερα την τηλεόρασή σου, δεν ξέρεις τι επίπεδο προστασία σου παρέχεται. Και πρέπει να υποθέσετε ότι δεν υπάρχει επίπεδο προστασία. Και νομίζω ότι αυτή η ειλικρίνεια είναι καλύτερη τελικά από το μία ψευδέστηση που μπορεί να δίνουμε στον καταναλωτή ε, ότι υπάρχει ένα είδο προστασία, ένα επίπεδο προστασία το οποίο τελικά δεν υπάρχει. Σίγουρα θα υπάρξει προσφορά, σίγουρα πολλοί α, ε, ε, καταναλωτές θέλουν καλύτερο επίπεδο α, ποιότητας. Αυτό βεβαίως το υποστηρίζουμε και νομίζω ότι είναι σημαντικό σημείο. Υπάρχουν κάποια καλά σημεία στην οδηγία με τα οποία μπορούμε να, να δουλέψουμε έτσι ώστε να υπάρχει καλή ποιότητα στις υπηρεσίες αυτές. Αλλά αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια εθελούσια βάση. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει ουσιαστικά αυτορύθμιση των παρόχων. Τη στιγμή που το προβλέψουμε εμείς πρέπει πάλι να το ελέγξουμε. Και πάλι εκεί μιλούμε για την εποπτεία. Επί της αρχής λοιπόν η βασική πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι να θέσουμε κριτήρια τα οποία αυτή την, ε, θα, προσφέρουν ε, την ε, δυνατότητα, θα, προσφέρουν ένα πλαίσιο, αλλά θα μπορούν να, να, να θεωρηθούν και από τους παρόχους ως εθελοντικά κριτήρια. Με την προϋπόθεση βεβαίως ότι όλα αυτά θα παρέχουν μια απαραίτητη ασφάλεια για τους καταναλωτές. Αυτό το σύστημα που λες εσύ, Πέτρα, στην έκθεσή σου για το, για το σύστημα με τα κίνητρα, έτσι ώστε και ο πάροχος να μπορεί να είναι πιο ψηλά στις καταχωρήσεις εφόσον παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες με το κατάλληλο επίπεδο προστασίας. Μπορούμε λοιπόν να διδεχτούμε την έκθεση. Το θέμα το, ε, της ισότητας όπλων είναι σημαντικό. Προφανώς δεν πρέπει να υπάρξει στεύρωση του ανταγωνισμού. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να είναι σαφές ότι στους καταναλωτές δεν πρέπει να δώσουμε ε, μια ιονή προστασία. Δεν τους κάνουμε καθόλου καλό. Μόνο όταν θα πληρούνται κάποια κριτήρια, μόνο τότε θα, μπορούμε, θα μπορούν οι πάροχοι να ε, εμφανίζονται πολύ, πιο, πολύ περισσότερο. Γιατί μετά θα πρέπει πάλι να περάσουμε σε επίπεδα ε, ελέγχου. Ο κύριο Κύρκοπ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη καταρχά. εκ μέρου τη κυρία Μακλάρκιν που δεν μπορεί να είναι παρούσα και μου ζήτησε να την αντικαταστήσω να μιλήσω για αυτό το θέμα το οποίο με ενδιαφέρει και εμένα προσωπικά ιδιαίτερα. Με Ενδιαφέραν πάντοτε τα μέσα μαζική ενημέρωση και με ενδιαφέρουν πολύ οι προτάσει τη εισηγητρίας. Πρώτα απ' όλα. Εν γέννη η έκθεση είναι καλή έρχεται ως προσθήκη της έκθεσης για τις οπτακουστικές υπηρεσίες και τη σχετική οδηγία. Και είναι πολύ σημαντικό νομίζω εμείς να εκμεταλλευτούμε για την κατάρτιση της έκθεσης αυτής της σχέσης συνδεδεμένη τηλεόραση. Να εκμεταλλευτούμε λοιπόν την ευκαιρία αυτή ώστε να επιστήσουμε του σε ορισμένα πράγματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ε, οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί οι κατάλληλοι, διότι μιλάμε για κάτι που εκφύσεως είναι παγκοσμιοποιημένο. Ο εξοπλισμός βέβαια για τη συνδεδεμένη τηλεόραση, την υπηρετική πλατφόρμα αυτή είναι κάτι που είναι κοινό σε αρκετές χώρες μελίδη μεταξύ αυτών και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά εδώ υπάρχει μια επανάσταση ως προς την ανάπτυξη λογισμικού, όχι μόνο για τη συνδεδεμένη τηλεόραση, αλλά και ευρύτερα. Υπάρχει μεγαλύτερη προσωποποίηση της τηλεόρασης. Όταν με ενδιαφέρε το θέμα πριν από κάποια χρόνια, η τηλεόραση αναπόφευκτα σχεδόν είχε να κάνει με την ε, συμμετοχή της κοινωνίας. Ε, βασιζόταν στην κοινωνία. Και όταν λέω κοινωνία μπορεί να είναι και μια πολύ ε, ολιγομελής, μια οικογένεια για παράδειγμα. Σήμερα όμως ε, με την... Όπως μου δείχνει ένας φίλος μου πρόσφατα, ε, την οθόνη της τηλεόρασης που την είχε βάλει στο ψυγείο του πάνω, στη, στην πόρτα Εντάξει, δεν ξέρω αν αυτό ήταν ένα τρόπο για να μην κάθεται αλλού με τα παιδιά του γυναίκα αλλά τέλο πάντων ε, είναι σημαντικό γιατί μπαίνει παντού μια οθόνη τη τηλεόραση και με τα κοινωνικά μέσα ενημέρωση βλέπουμε να συντελείται μια τεράστια αλλαγή. Και βέβαια και οι διαφημιστέ οι οποίοι εκμεταλλεύονται τα πάντα, ό,τι βρίσκεται από την άλλη πλευρά τη οθόνη. Είναι λοιπόν ε, συναρπαστική αυτή η καινοτομία τη ευρωπαϊκή τηλεόραση. Ε, εξελίσσεται συνεχώ η πλατφόρμα, αλλά θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μα και του κινδύνου αλλά και τη διαφήμιση. Και έχουμε να κάνουμε κανόνες ε, δικαιωμάτων δημιουργού, copyright, έχουμε να κάνουμε με θέματα προστασίας, ιδίως των παιδιών. Η Έμα μου ζήτησε να σας ε, επισημάνω ότι θα την ενδιαφέρει ιδιαίτερα να γίνεται περισσότερη μνήα εδώ στην προστασία των ανηλίκων, διότι νομίζω ότι και πάλι για του λόγου που σας προανέφερα, η νεολαία σήμερα επηρεάζεται πολύ περισσότερο από ό,τι παλαιότερα από αυτό που βλέπεις στην οθόνη. Κυρίως γιατί κάθε μπροστά από την οθόνη μόνοι τους ε, κάθονται οι νέοι, όχι ε, με την επίβλεψη κάποιου μεγαλύτερου. Επίσης, ε, κάτι άλλο που είναι σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι για να απολαύσει κανείς την υπηρετική τηλεόραση και άλλες τέτοιες τεχνολογίες θα πρέπει να έχει μεγάλη ταχύτητα δίκτυο. Ξέρουμε όμω ότι υπάρχουν περιοχέ με περιορισμένη διαδικτυακή υποδομή. Κάποιε χώρε σημειώνουν πρόοδο και αυτό είναι καλό. Καλό όχι μόνο για την κοινωνική χρήση, αλλά και για την επιχειρηματική χρήση των εξέλιξεων αυτών. Άρα αυτό πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι καλό και για την Ευρώπη. Νομίζω όμω ότι θα πρέπει στην έκθεση να τονιστεί περισσότερο η ανάγκη τη μεγαλύτερη διαδικτυακή ταχύτητα. Εν τέλει, ε, να πω ότι φυσικά και θα συνεργαστούμε απόλυτα με την εισηγήτρια. Η κυρία Μακλάρκιν τους επόμενους μήνες θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα. Και να πω και κάτι ακόμη, ότι το πρόβλημα είναι ότι οι νομοθέτες κινούμαστε με πολύ μικρότερη ταχύτητα και δεν έχουμε πάντοτε και τη σωστή απάντηση σε όλα. Στην προκειμένη περίπτωση όμως νομίζω ότι θα πρέπει να μην μείνουμε πίσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λέει ο πρόεδρο, ο κύριο Καβαντά. Συγγνώμη, κύριε Καβαντά, δεν σα είδα πριν. Κύριο Καβαντά. Σα ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Γιατί είδατε ότι έκανα χειρονομίε. Ε, Δυστυχώ, ε, επειδή μα ε, χωρί μια μεγάλη απόσταση τη γραμματεία, ήμουν αόρατο για τη γραμματεία. Τέλο πάντων, θέλω να σα ευχαριστήσω, Πέτρα, για την έκθεσή σα, όπω και οι προλήσατε συναδελφοί μου. Και για να μην φλιαρώ, ε, ίσως 6 Μαρτίου στην επίδειξη που θα κάνετε στο του Μονάχου θα δούμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται και φαντάζομαι ότι αυτό θα είναι και η απαρχή γιατί είναι η αρχή αυτής της περιπέτειας και δεν μπορούμε να υπολογίσουμε όλες τις συνέπειες ε, που θα έχει αυτό. Πριν από δύο μήνες περίπου η ομάδα μου και εγώ για μια μέρα κάναμε ακριβώς, ε, είχαμε την ίδια αυτή εμπειρία διαφόρους, με διάφορα, διάφορα είδη βρετικής τηλεόρασης, ήρθαμε σε, σε επαφή και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθεί κανείς τις επιπτώσεις αυτού που τώρα εξετάζουμε. Και οι επιπτώσεις, ήδη αρχίσουμε κάπως να τις διαβλέπουμε, ενδεχομένως να υπάρξουν ε, ε, κάποια ολιστήματα, εκτροπές, είπατε και εσείς αγαπητοί συνάδελφε, και σίγουρα πρέπει να σκεφτούμε, να σκεφτούμε πώς θα οργανώσουμε τα πράγματα, το είπε και ο Κύρκο, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι σήμερα είμαστε ε, στην αρχή, στο εμβριο, εμβριακό ακόμη στάδιο αυτής της ευρετικής τηλεόρασης και δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τα πράγματα ε, εξαντλητικά, διεξοδικά. Καταλαβαίνω ότι πολλά διακυβεύονται, καταλαβαίνω και τις ανησυχίες σας, αλλά θεωρώ ότι θα ήταν λίγο πρόημο να μιλήσουμε για μια άρδιν ε, αναθεώρηση της οδηγίας ε, SMA. Είμαστε στην αρχή ακόμη. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε ή δεν πορελέψαμε και τώρα, αλλά και στο μέλλον θα μπορούμε να δούμε ακριβώ τι ε, εξέλιξη μπορεί να υπάρξει με αυτή την τεχνολογία. πρέπει να μπορούμε να είμαστε ταυτόχρονα ως συνομοθέτες ε, σόφρονες, συνετοί και ταυτόχρονα βέβαια να λάβουμε και τις ευθύνες. Τι θα πει αυτό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών ομήλων για τις επενδύσεις. Με ενδεχομένη νοσμόνη εξαίρεση την Γερμανία που η δημόσια όμιλη είναι πολύ ισχυρή, το ίδιο δεν ισχύει στι άλλε χώρε. Και αυτό δεν είναι φυσιολογικό γιατί επηρεάζει το περιεχόμενο βέβαια. Δεύτερη αρχή που πρέπει να σεβαστούμε είναι η ελευθερία. Υπογραμμίσατε κι εσεί, Πέτρα, το θέμα αυτό. Νομίζω ότι δεν αμφισβητείται από κανέναν και είναι και κάτι καλό. Αλλά ούτε και εδώ, ούτε και στις χώρες ε, ακούω πολλά πράγματα ε, για το τρίτο πολύ σημαντικό θέμα που είναι η ευθύνη. Προστασία των ανηλίκων. Θα ήθελε κανείς από εσάς να εκτίθεται τα παιδιά του σε ό,τι περιεχόμενο ε, διακινείται μέσω του διαδικτύου. και βέβαια μπορεί κανείς να είναι ευλαβικά προσιλωμένος στην ελευθερία, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει αυτό να οδηγήσει σε ανευθυνότητα ή και σε μία ε, συνενοχή στην τρέλα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μία, ένα συγκερασμός όλων αυτό. Τι θέλουμε. Θέλουμε διαφημίσεις που κάπου να διακόπτονται από πρόγραμμα ε, ή το αντίστροφο, να έχουμε προγράμματα που μπορεί να διακόπτονται που και από διαφημίσεις και σίγουρα τα 12 λεπτά δεν τα σέβονται όλες ε, οι χώρες παρότι αυτό το έχει ρυθμίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είχα να πω για το πρώτο σημείο. Θα ήθελα όμως να κάνω και κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με τους οπτικοακουστικούς φορείς, ε, τους επιδραμικούς που ε, ε, δεν έχουν τις ίδιες δεν, δεν έχουν τις υποχρεώσεις με τους κλασικούς παραδοσιακούς οπτικοακουστικούς φορείς. Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε όλους τους κανόνες να τους διαγράψουμε. Μην είμαστε τόσο απρόσεκτοι, να μην αφήσουμε χωρίς πλαίσιο αυτούς τους φορείς. Η οικονομία επενδύσεων είναι ο καθορισμός του πλαισίου δεν καταργεί την ελευθερία. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο που στηρίζεται και στις τεχνολογίες για να αυξήσει την, αποτελεσματικότητα, το profiling των καταναλωτών κτλ. Πολιοθωνικές, στρατηγικές που θα κάνουν θράψη και ούτω, και ε, ούτω καθεξής. Ε, δημιουργούν και άλλα ζητήματα, προστασία ιδιωτικής ζωής και βέβαια σε καμία περίπτωση ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής ε, δεν θα πρέπει να διαχωρίζεται απόλυτα από την ανάγκη για προστασία. Και δεν είναι φυσιολογικό η ένωμη τάξη, η δημόσια τάξη, να μην ε, λαμβάνεται υπόψη σε αυτό το θέμα. Φυσικά η ευθύνη και η ευθύνη ε, των ε, αρχισυντακτών, της σύνταξη είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό και της επιμέλειας, διότι δεν μιλάμε για εμπορικά προϊόντα, Μπορεί να υπάρχει και εμπορική δραστηριότητα, αλλά αυτό είναι όλο. Θα σας προτείνω πάντως, αγαπητοί συνάδελφοι, τροπολογίες για τα διάφορα σημεία και φαντάζομαι ότι στην πρώτη έκθεση, στο, στο πρώτο σχέδιο, το οποίο είναι πολλά υποσχόμενο, θα μπορέσουμε να συζητήσουμε διεξοδικότερα. Σας ευχαριστώ πάντως. Σας ευχαριστώ. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είστε εδώ. Ωραία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαστε ιδιαίτερα. Νομίζω ότι είχα την ευκαιρία να σας το πω και προσωπικώς, ε, κυρίως ε, στην εισηγήτρια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ ικανοποιημένη ε, για το ενδιαφέρον που δημιουργεί το συγκεκριμένο ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι πιστεύουμε ότι αξίζει αυτό το ενδιαφέρον που, που δείχνεται. Διαμαρτύρεστε ότι έχετε περιορισμένο αριθμό λέξεων, παρόλα αυτά εμεί θεωρούμε ότι λέτε πολλά πράγματα στο λίγο χώρο ε, τον οποίο έχετε στη διάθεσή σα για την έκθεση. Πολλοί από εσά φαίνεται να έχετε ήδη καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πρέπει να αλλάξουμε την οδηγία για τις υπηρεσίες των οπτικοακουστικών μέσων. Δεν συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως γνωρίζετε αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία της αξιολόγησης και η πράσινη βίβλος είναι το εργαλείο που χρησιμοποιούμε προς αυτό το σκοπό και νομίζω ότι η κυρία Καμερβέλη πολύ σωστά είπε ότι αυτή δεν είναι μια ε, οποιαδήποτε οδηγία, είναι μια οδηγία η οποία προστατεύει αξίες και αποφασίστηκε από τον νομοθέτη ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη οδηγία για αυτά τα ζητήματα και επομένως θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ε, είναι νωρίς ακόμα, είμαστε στα Σπάργανα γνωρίζουμε ότι περισσότεροι ξημών έχουμε μία ε, συνδεδεμένη τηλεόραση, αλλά ελάχιστοι δυστυχώς τη χρησιμοποιούν ε, όπως πρέπει. Τα ποσοστά λοιπόν είναι πολύ χαμηλά ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στρατηγική λοιπόν που αποφάσισε να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι δεν θα καθίσουμε με σταυρωμένα χέρια να δούμε τι θα συμβεί και να βρεθούμε με στη συνέχεια πρώτα τελεσμένου όπως ε, είπε και η κυρία Κάμερβεν. Θα προσπαθήσουμε να ε, ανοίξουμε τη συζήτηση, να γίνει ε, διαβούλευση, να διαπιστώσουμε τι συμβαίνει και κατόπιν να αποφασίσουμε. Θεωρούμε ότι η συζήτηση αυτή είναι πολύ χρήσιμη για αυτό που κάνουμε, ιδιαίτερα χρήσιμη. Η έκθεση είναι πολλά υποσχόμενη όπως ε, αναφέρθηκε και προηγουμένως. Κατά τα λοιπά, όπως γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συζητούμε το έγγραφο με τους συναδέλφους από τις άλλες γενικές διευθύνσεις. Επομένως, είναι πολύ νωρίς ε, για να σας πω τι ακριβώς θα λέει η έκθεση. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι το πεδίο εφαρμογής θα καλύπτει όπως είπατε και κάποιοι από εσά, όπως η κυρία και κινητές συσκευέ, όχι μόνο τη συνδεδεμένη τηλεόραση και κατά τα λοιπά, όλα τα θέματα τα οποία συζητώνται, τα περισσότερα εξ αυτών, ε, έχουμε πρόθεση να τα καλύψουμε. Και θα θέσουμε ερωτήσεις και θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια ισορροπία μεταξύ ευελιξίας, προστασίας των καταναλωτών και πολλών άλλων αξιών που προσπαθεί να προασπίσει η συγκεκριμένη οδηγία. Αυτά λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, συζήτηση αυτή. Εγώ ευχαριστώ. Πέτρα, σύντομα. Äh, Θα είμαι σύντομη, Πρόεδρε. Ο Jean-Marie έφυγε. Αλλά ακριβώ ήθελα να του πω ότι δεν είναι νωρί να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό και να το συζητήσουμε. Καθόλου νωρί δεν είναι να δούμε ποια είναι η κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα όρο, καλό, σωστό συντονισμό για τα ΜΜΕ για το μέλλον. Ε, η Κομισιόν όλο αναβάλει την έκδοση της Πράσινης Βίβλου της όμως. Ε, θα ερχόταν το φθινόπωρο. Τώρα η προθεσμία είναι τον Απρίλιο. Ναι, αλλά αυτό μας κοστίζει πολύτιμο χρόνο, γιατί έχουμε και μια διαδικασία διαβούλευσης και πρέπει να πάρουμε και μια θέση. Και μας κοστίζει χρόνο, γιατί κοστίζει χρόνο στην νομοθετική διαδικασία. Πρέπει να απαντήσουμε, να αντιδράσουμε άμεσα. Να μην δημιουργηθούν δηλαδή τελεσμένα τα οποία να μην μπορούμε μετά να τα αναστρέψουμε εμεί ω πολιτικοί ή να βρεθούμε πάλι σε μια κατάσταση που θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γι' αυτό ζητώ να ε, βιαστούμε λιγάκι όταν μιλούμε για τέτοια πράγματα, για τέτοια θέματα πολιτικής, ε, για τα ΜΜΕ. Για την κυρία Χίρς, ε, ρυθμισμένη αυτορύθμιση. Δεν θέλω να τα αφήσουμε όλα σε αυτό το τομέα της ρυθμισμένης αυτορύθμισης, αλλά όταν κάποιο έχει ε, έτσι, προνόμια, ε, αυτό τα έχει λόγω κάποιων προϋποθέσεων τις οποίες πληρεί. Πρέπει πρώτα να τις πληρεί και μετά θα μπορεί κάποιος να ελέγχει αν όντω όλα όσα προβλέπονται τηρούνται. Τι κάνει δηλαδή ο ε, ελεγκτής του δημόσια, της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Ε, αυτό όλα αυτά μπορούν να ελεγχθούν. Δεν είναι δηλαδή ότι εγώ μια φορά πήρα μια πιστοποίηση και μπορεί να ισχύει για πάντα. Όχι. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται μόνο αυτορύθμιση, χρειάζεται ρυθμισμένη αυτορύθμιση. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε βεβαίω για τα παιδιά, για την προστασία των παιδιών κτλ. Φυσικά και θα το κάνουμε, αλλά εξακολουθεί να είναι αυτό ρύθμιση των ΜΜΕ, εξακολουθούν να είναι κανόνε, οι κανόνε πρέπει να πληρούνται και βεβαίω αυτό πρέπει να, εξ, ε, ε, εξετάζεται. Το θέμα τη προστασία στο διαδίκτυο για τα παιδιά είναι θέμα σημαντικό. Ε, δεν μπορούμε να ελέγξουμε το διαδίκτυο, προφανώ και ούτε θέλουμε, αλλά πρέπει να δούμε πώ μπορούμε με κάποιο λογικό τρόπο να το διαχειριστούμε και πώ μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτά τα προνόμια δεν θα τυχάνουν και οποιασδήποτε κατάχρηση. Και αυτό είναι σημαντικό. Κατά τα λοιπά, χαίρομαι για τι τροπολογίες σα, θα τι περιμένω. Χαίρομαι που θα κάνουμε και άλλε ωραίε συζητήσει σαν τη σημερινή, έτσι ώστε να καταλήξουμε τελικά στην ψήφιση τη ε, οδηγία. Σα ευχαριστώ για τι παρεμβάσει σα. Εγώ ευχαριστώ. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Έτσι ώστε να εμπλουτιστεί κι άλλο η έκθεση. Είναι λίγο περίεργο να υποβάλει κανεί βέβαια τροπολογία στη δική σου έκθεση, αλλά 5η, 7 Μαρτίου, του τρέχοντος έχετε την ε, δυνατότητα να υποβάλλετε τις, ε, τις τροπολογίες σας. Θέλουμε να είμαστε λίγο πιο γρήγοροι από την Κομισιόν. Η κυρία Πέτρα λέει πάντα είμαστε πιο γρήγοροι από την Κομισιόν. Αν σκεφτείτε πόσο χρόνο έχουμε δαπανίσει για να, να, να, να συλλάβουμε το θέμα της διαφήμισης και να το συμπεριλάβουμε σε μία α, έκθεση, πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον. Φυσικά πάντα μπορούμε να αποδειχθούμε λιγάκι πιο έξυπνοι. Ε, λοιπόν, Πέρα τη ε, ε, συνεδρίαση. Θα τα πούμε αύριο στις 9 το πρωί για να ψηφίσουμε. Όποιο δεν είναι αύριο εδώ, παρακαλώ στείλτε εκπροσώπους σα, αντιπροσώπους. Τώρα, έχουμε τους συντονιστές. Όλοι οι υπόλοιποι παρακαλώ να αποχωρήσουν από αυτό το απέσιο κρύο δωμάτιο και να βρουν ένα, μια πιο ωραία αίθουσα. Two minutes forward.